Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρία τη Επιτροπής Προϋπολογισμών και θα ήθελα να καλωσορίσω στη συνεδρίασή μας τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Ο πρόεδρος δεν έχει έρθει ακόμη, δεν μπόρεσε να έρθει. Θα συζητήσουμε την διορθωτική επιστολή για τον προϋπολογισμό του 2015 και στη συζήτηση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το λόγο και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Πολύ σημαντική σημερινή μας συνεδρίαση, γιατί είμαστε παραμονές της συνδιαλλαγής για τον διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2014 και το σχέδιο προϋπολογισμού του 2015. Καταρχήν, συμφωνούμε με την ημερήσια διάταξη. Μπορούμε να την εγκρίνουμε. Έχετε λίγα αντίτυπα των εγγράφων, γιατί προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κοινοβούλιο χωρίς χαρτί. Τα περισσότερα και τα πιο ογκώδη έγγραφα μπορείτε να τα λάβετε με ηλεκτρονική μορφή. Καταρχήν να σας ενημερώσω για τις αποφάσεις των συντονιστών στη συνεδρίαση της 22ης Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά την ε, δυνατότητα υποβολή σχεδίου γνωμοδότησης ε, για την έκθεση εκών και απασχόλησης για το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη μέχρι τώρα πρακτική και να συντάξουμε μία και μόνο γνωμοδότηση επί της ε, εκθέσεως της ΕΚΟΝ. Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια του τριμερούς διαλόγου της 15ης Οκτωβρίου, οι συντονιστές επιβεβαίωσαν το στρατηγικό τους όραμα και θεωρούν ότι η συνδιαλλαγή θα πρέπει να ασχοληθεί πρώτα με τα σχέδια διορθωτικού προπολογισμού του 2014 πριν υπησέλθει στην εξέταση του προπολογισμού του 2015. Σε ό,τι αφορά τα σχέδια ε, διορθωτικών προπολογισμών 2 έως 7, οι συντονιστές συμφώνησαν να παραμείνουν τα σχέδια αυτά ενιαία σε ένα πακέτο, σε ένα ενιαίο πακέτο, αδιέρετο. Και σε ό,τι αφορά τα σημεία 3 ως 7, θα πρέπει να ψηφίσουμε σε μια ενδεικτική ψηφοφορία επί των εκθέσεων του κ. Ζεράρντε πρέ. Για τα εκρεμή θέματα που αφορούν τους προϋπολογισμούς 2014 και 2015, απόφαση ποιήσης του Ταμείου Αλληλεγγύης, η πρόταση της χρήσης του μέσου ευελιξίας και του περιθωρίου για τα απρόπτα περιστατικά, της απρόπτες ανάγκες. Οι συντονιστές ε, θεώρησαν ότι καλό θα ήταν να ψηφίσουμε για τα θέματα αυτά μετά την ε, ολοκλήρωση της συζήτησης ε, στη συνδιαλλαγή. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, αν ευοδοθεί η συνδιαλλαγή στις 14 Νοεμβρίου, προβλέπει εξέταση στις 20 Νοεμβρίου. Αυτό είναι το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα σε περίπτωση που τελεσφορήσει η συνδιαλλαγή. Αυτά ως προς ανακοινώσεις. Τώρα να επισέλθουμε στη διορθωτική επιστολή για τον προπολογισμό του 2015. Και ευχαριστώ και την κυρία Καλβίνιο που ήρθε και θα την παρακαλούσα να μας παρουσιάσει αυτή την διορθωτική επιστολή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε αυτή τη διορθωτική επιστολή. Ως συνήθως και πριν την έναρξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής όπως είπατε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη διορθωτική της επιστολή προκειμένου να ληφθεί υπόψη να η υπόψη τελευταίες εξελίξεις ως προς την εφαρμογή της κοινή γεωργικής πολιτικής. Δεδομένων των ε, γνωστών σε σας ε, περιστάσεων και ιδιαίτερα της, ε, του περιορισμένου ποσού των πιστώσεων πληρωμών. Φέτος ε, στην διορθωτική μα επιστολή θετήσαμε μια πολύ στεναρή και αυστηρή προσέγγιση προκειμένου να βρούμε ποιο είναι ο πιο αποτελεσματικός και αποδοτικό τρόπο για να καλύψουμε τι ανάγκε τη κοινή αγροτική πολιτική ε, από άποψη δημοσιονομική εννοώ. Η πρόταση δημιούργησε πολλά ερωτηματικά και Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων ε, ότι, για το γεγονό ότι προσκαλέσατε και τα μέλη τη Επιτροπή ε, Γεωργία στη συνεδρία κατά την οποία θα γίνει η παρουσίαση αυτή τη διορθωτική επιστολή. Οι δαπάνε ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου, Γεωργικού Ταμείου Αγγίσεων χρηματοδοτούν, το καταμείο αυτό χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού αλλά και από σημαντικό ποσό προσημειωμένων πιστώσεων που προκύπτουν από διορθώσει σε σχέση με τι δαπάνε του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, εκαθάριση λογαριασμών, κάποιε παρατυπίε και τις συνεισφορές των ε, παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων. Επίσης λαμβάνονται υπόψη τα πλεονάσματα της ε, τρέχουσας δημοσιονομικής χρήσης του 2014 και της αυτόματης μεταφοράς τους ε, στον επόμενο προϋπολογισμό. Οπότε αυτό το μεγάλο ποσοστό αναδιατεταγμένων αναδιατεταγμένο πιστώσεων μας επιτρέπει να κάνουμε κάποιες διορθώσεις στον προηγούμενο προπολογισμό της Άνοιξης και τα οι πιστώσει ε, τη κοινή γεωργική πολιτική, ε, τα σχετικά κονδύλια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων. Οπότε στην πράξη τα έσοδα αυτά προσθέτονται στο Ανώτατο Ταμείο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου. Θα ήθελα να τονίσω ότι λαμβάνουμε υπόψη ότι τα έσοδα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη γεωργία και επίσης αποτελούν νέα κονδύλια της κοινή γεωργικής πολιτικής. Επιπλέον το αρνητά του αρίου που προβλέπεται στο προϋπολογισμό διορθωτική στην διορθωτική επιστολή έχουν αυξηθεί τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων κατά 17 εκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει στον πίνακα που βλέπετε. Αυτό ανταποκρίνεται στι ε, προβλεπόμενε ανάγκε δεδομένων και των επιπλέον εσόδων. Τα έσοδα αυτά θα αυξηθούν κατά 465 εκατομμύρια σε σύγκριση με τι αρχικέ προβλέψει που είχαμε κάνει την άνοιξη του τρέχοντο έτου. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι αυτά τα έσοδα προβλέπονται στον ε, συγκεκριτικό προϋπολογισμό και έχουμε με βάση αυτό το ποσό έχουμε μείωση κατά 448 εκατομμύρια ευρώ στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο. Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων παραμένουν στην κατηγορία 2, οπότε αυξάνεται το περιθώριο κατά 734 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε οι αναλήψεις υποχρεώσεων προβλέπονται για την κάλυψη των γεωργικών ε, δαπανών. Θα ήθελα να επιμένω σε τρία σημεία. Δεν αφαιρούμε κονδύλια από τη γεωργία. Το αντίθετο, έχουμε περισσότερα κονδύλια για το γεωργικό ταμείο μετά την διορθωτική επιστολή από ό,τι είχαμε πριν τη διορθωτική επιστολή. Οπότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα νέα ποσά και έτσι διαπιστώνουμε ότι έχουμε περισσότερα κονδύλια για την κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης δεν αφορούμε κάποια έσοδα για να χρηματοδοτήσουμε μη γεωργικές δαπάνες. Αυτό τους άλλως δεν ε, προβλέπεται και νομικά. Και οι εισφορές από τα γαλακτοκομικά δεν έχουν προσημειωθεί για, τα, για συγκεκριμένα μέτρα, αλλά χρηματοδοτούν τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου. Η επόμενη διαφάνεια αναφέρεται σε ένα ειδικό θέμα θετινό που, λέει που προβλέπει την χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων για τη διόρθωση των ζημιών από το ρωσικό εμπάργο. Όπως ξέρετε, ε, η γεωρική χρήση φτάνει μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, οπότε τα επιπλέον έξοδα επιβαρύνουν την επόμενη δημοσιονομική χρονιά. Οι προβλεπόμενες ανάγκες για φέτος, ε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κρίση που δημιουργήθηκε από το ρωσικό εμπάργο, είναι 324 εκατομμύρια για τα προκυβευτικά και 20 εκατομμύρια για τον γαλακτοκομικό τομέα. Αυτό προβλέπεται στον προϋπολογισμό. Το ρωσικό εμπάργο όμως είναι καλή περίπτωση για να δούμε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Όταν ξεκίνησε η κρίση στα μέσα του καλοκαιριού, ενώ έχουμε τα έξοδα μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, ε, οι δαπάνε αυτές δεν επιβαρύνουν τον τρέχοντα προϋπολογισμό, αλλά θα πρέπει να μετακυληθούν στον επόμενο προϋπολογισμό, το 2015. Γι' αυτό και το αποθεματικό της κρίσης για το 2014 δεν χρησιμοποιήθηκε, αλλά περνάει στο 2015 και επιπλέον έχουμε 450 επιπλέον εκατομμύρια που αφαιρούμε από τι άμεσε ενισχύσει με βάση την εφαρμογή τη δημοσιονομική πειθαρχία. Οπότε, το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση που λαμβάνει η χώρα στο δεύτερο εξάμεινο του έτους. Μπορεί το αποθεματικό κρίση να χρησιμοποιηθεί για μια κρίση που λαμβάνει η χώρα στο δεύτερο εξάμεινο. Δηλαδή, θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τη χρήση του αποθεματικού μόνο για το πρώτο εξάμεινο. Όχι βέβαια. Αυτή την κατάσταση χρειάστηκε να λάβουμε υπόψη όταν συντάξαμε την διορθωτική επιστολή. Πώς όμως θα κινητοποιήσουμε το αποθεματικό της κρίσης. Το πρώτο βήμα είναι να αξιολογήσουμε τις τρέχουσες ανάγκες με βάση την εφαρμογή των μέτρων. Το δεύτερο βήμα είναι να δούμε αν υπάρχουν πιστώσεις διαθέσιμες στις δημοσιονομικές γραμμές. Αν είναι ανεπαρκής θα πρέπει να δούμε άλλα έσοδα πέραν των προσημειωμένων και επίσης είναι πολύ πιθανό φέτος να του χρόνου να έχουμε περισσότερα έσοδα δεδομένων των συζητήσεων που έχουμε με κράτη-μέλη για τις διορθώσεις. Και τέλος, αφού εξαντλήσουμε όλες τις ε, προηγούμενες εναλλακτικέ, θα προτείνουμε μεταφορά με βάση το αποθεματικό και με βάση το άρθρο 22. Για το πρώτο βήμα για να σας δείξω πώς λειτουργεί η διαδικασία. Έχουμε ήδη κάποια νέα σχετικά. Με βάση τις τελευταίες ε, κοινοποίησεις που έγιναν από τα κράτη-μέλη για το πρώτο έκτακτο πακέτο για τα προκυπευτικά, μόνο 30% προκύπτει από τα 37,3 εκατομμύρια, από τις αρχικές προβλέψεις των 125 εκατομμύριων, αφορούν επιλέξιμες δαπάνες. Οπότε επιβεβαιώνεται η εντύπωση που είχαμε ότι το πρώτο κύμα ε, συζητήσεων ήταν υπερτιμημένο. Οπότε ο προπολογισμό που είχαμε προβλέψει για την αντιμετώπιση της κρίσης ήταν διωγγωμένος, γιατί τελικά οι ανάγκες θα είναι χαμηλότερες από ό,τι είχαμε αναμείνει. Τώρα για την ιδιωτική αποθεματοποίηση του τυριού, το ίδιο ισχύει. Το σύστημα σταμάτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί οι περισσότερες αιτήσει έγιναν από παραγωγούς που δεν ε, εξήγαν προς τη Ρωσία. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και οι πραγματικές ζημίες ε, του ρωσικού εμπάργου. Μετά λοιπόν τα τελευταία στοιχεία για τα εφαρμοστέα μέτρα ε, θεωρούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εξαντλήσουμε καν το αποθεματικό της κρίσης το 2015. Οι νέες προβλέψεις για το εναπομείνα ποσό είναι 180 περίπου εκατομμύρια αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα 88,7 εκατομμύρια που είχαμε όταν κατά προτείναμε τον, την διορθωτική επιστολή και βρισκόμαστε ακόμη στο πρώτο βήμα της διαδικασίας αυτής. Η τελευταία διαφάνεια αφορά και πάλι το αποθεματικό της κρίσης γιατί αναφέραμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί αυτό το αποθεματικό και είχαμε κάποιες αντιρρήσεις είναι το έσχατο μέσο το αποθεματικό της κρίσης. Ήδη περιλαμβάνεται στο 2015 για ποσό 133 εκατομμυρίων και ανεξάρτητα από τη χρήση του, το αποθεματικό αυτό για τις απρόβλεπτες ανάγκες ε, προβλέφθηκε στην αρχή του έτους για τη μείωση των άμεσων ενισχύσεων και με την πραγματική εφαρμογή του Γεωργικού Ταμείου θα κρίνουμε κατά πόσο θα, θα χρησιμοποιήσουμε και για ποια ποσά το αποθεματικό των απρόβλεπτων αναγκών. Η χρήση του θα, ε, θα εξαρτηθεί από την πραγματική εφαρμογή των κονδυλίων του Γεωργικού Ταμείου. Οπότε δεν είναι σωστό να λέμε ότι αυτή τη στιγμή οι γεωργοί πληρώνουν τα σπασμένα των μέτρων της κρίσης. Και επειδή προέκυψαν αντιδράσεις όταν προτείναμε την πιθανότητα της χρήσης του εναλλακτικού κρίσης, να σας πω ότι το 2015 έχουμε πρώτη φορά τη δημοσιονομική πειθαρχία. Το μέτρο αυτό υπήρχε από το 2006 θεωρητικά, αλλά φαίνεται ότι για πρώτη φορά ε, ο κόσμος διαπιστώνει ότι το εφαρμόζουμε και στην πράξη. Και ό,τι είχαμε τα πρώτα έγγραφα για το 2014, τα κακά μαντάτα για την δημοσιονομική πειθαρχία αναφερόταν κυρίως στη Γεωργία με πολύ αρνητικά σχόλια. Προς τα τέλη του 2015 όμως ε, θα έχουμε μια κατάσταση στο Γεωργικό Ταμείο που θα προβλέπει επιστροφή του συνολικού ποσού της, της δημοσιονομικής πειθαρχίας κατά την αρχή του 2015. Και αυτά τα καλά μανδάτα τα αναφέρουμε στην διορθωτική επιστολή για το 2015. Στην αρχή είχαμε διαμαρτυρίες και αρνητικές αντιδράσεις και τώρα βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο του ποσού θα επιστραφεί. Τώρα, τι προτείνουμε με τις πιστώσεις που θα απελευθερωθούν με το επιπλέον έσοδα που θα κατανεμηθούν. Προτείνουμε αναδιάταξη των πληρωμών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες άλλων τμήματων του προϋπολογισμού. Τους τελευταίους μήνες είχαμε πολλές περιπτώσεις για να ε, εξετάσουμε την δύσκολη θέση με τις πιστώσεις πληρωμών και είχαμε και τη διοργανική παρουσίαση εδώ το Σεπτέμβριο Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη συνολική μεταφορά για την αναδιάταξη των πιστώσεων πληρωμών στα τμήματα του προπολογισμού που ε, παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Φέτος είναι χαμηλότερη η μεταφορά, είναι μόνο 175 εκατομμύρια. Δεν μας εκπλήσει αυτό, γιατί η κατάσταση στον προπολογισμό είναι πραγματικά πολύ σφιχτή. Ο Πρόεδρος διακόπτει. Μήπω μπορείτε να επιβραδύνετε λίγο το ρυθμό σας, γιατί πραγματικά μιλάτε σαν μετραλιογόλο. Ναι, ναι, ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Ναι, όντω μιλάω αρκετά γρήγορα. Τώρα, τι θα, τι θα κάνουμε με τις πιστώσεις πληρωμών που θα απελευθερωθούν χάρη στα έσοδα ειδικού προορισμού που έχουμε εντοπίσει. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν είναι να ανακατανύμουμε αυτές τις πιστώσεις πληρωμών στις ε, δημοσιονομικές γραμμές που παρουσιάζουν μεγαλύτερες ανάγκες. Θα, θυμάτε, θα θυμάστε ότι ο Επίτροπος Ντομινίκ σας παρουσίασε την δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στο φετινό προϋπολογισμό. Εξαιτίας τη μείωση των ανωτάτων ορίων του νέου Γεωργικού Ταμείου, αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες σε πολλές δημοσιονομικές γραμμές που έχουν ήδη εξαντληθεί και έτσι εξηγείται ε, το μικρό μέγεθος της ε, συνολικής μεταφοράς που είναι μόνο 175 εκατομμύρια. Είναι πραγματικά ιστορικά από τα χαμηλότερα ποσά. Και πιστώσεις πληρωμών που θα χρειαστούν για την, για την ανακατανομή είναι πολύ λίγες. Γι' αυτό στην διορθωτική επιστολή προτείνουμε αναδιάταξη ε, της τάξης 448 εκατομμυρίων ευρώ για να αποφύγουμε τόκους περιμερίες και να μειώσουμε τον αυξανόμενο, το αυξανόμενο κόστος των ε, οπισθοβαρών καταβολών. Βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια τις προτάσεις για τα προγράμματα που θα ενισχυθούν για το 2015 μέσω της αναδιάταξης πιστώσεων πληρωμών που θα προέλθουν από τον τομέα 2, από την κατηγορία 2 το, ο τομέας 1α θα απορροφήσει 240 εκατομμύρια, πάνω από τα μισά. Επίσης, ενεργειακά προγράμματα ε, που έχουν ε, πολλά, πολλά τιμολόγια που θα πρέπει να πληρωθούν. Θέλουμε να αποφύγουμε ε, να πληρώσουμε πολλού τόκου υπερημερίε. Έχουμε και το κλείσιμο του 7ου ερευνητικού προγράμματο πλαισίου και εκεί θα περιμένουμε πολλού λογαριασμού. Έχουμε τον ορίζοντα 2020, επίσης ε, πολλά, πολλούς ανεξόφλητους λογαριασμούς, οπότε τα περισσότερα κονδύλια θα πάνε στο 1α. Τώρα, στο 1β έχουμε 51 εκατομμύρια, θέλουμε να ολοκληρώσουμε τα περιβαλλοντικά προγράμματα, Life Sin, Επίσης θέλουμε να αποφύγουμε την καταβολή τόκων υπερημερίας και θέλουμε να ολοκληρώσουμε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας στον τομέα 2. Τώρα, επειδή έχουμε όλο και περισσότερες οπισθοβαρείς πληρωμές, έχουμε πρόβλημα στον τίτλο 4 και για την αναπτυξιακή συνεργασία και για την πολιτική γειτονία. Εκεί θέλουμε να μειώσουμε τον αυξανόμενο όγκο των ανεξόφλητων λογαριασμών. Οπότε είδατε πώς θα ανακατανύμουμε τις πιστώσεις πληρωμών στις ε, ε, στους συγκεκριμένους τομείς 1α, 2 και 4. Και περνάω στην τελευταία διαφάνεια με τα συμπεράσματα, μου επιτρέπετε. Συγγνώμη. Δεν είχα τσεχική διερμηνία. Καλά τα αγγλικά, αλλά γιατί δεν είχαμε τσεχική διερμηνία. Thank, thank you very much. Oui. Et... Bien. L'avez-vous... It's okay. Εντάξει τώρα, λύθηκε το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Και καλό θα ήταν να συνεχίσετε σε αυτό το πιο ήπιο ρυθμό. Ναι, φτάνουμε σιγά σιγά στα συμπεράσματα. Και πραγματικά ζητώ συγγνώμη γιατί από τεχνική άποψη είναι από τα πιο περίπλοκα τμήματα του προπολογισμού. και είναι δύσκολη και τεχνική ορολογία που χρησιμοποιώ. Είναι λογικό να μην μπορούν να με προλάβουν οι διερμηνείς όταν μιλάω γρήγορα. Φτάνουμε λοιπόν στα συμπεράσματα και ελπίζω από την παρουσίαση να ε, αντιληφθήκατε γιατί προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρώτη διορθωτική επιστολή και το 2015. Λοιπόν, πρώτο συμπέρασμα. Η διορθωτική προπολογισμή αυξάνει τα κονδύλια του Γεωργικού Ταμείου σε σχέση με, τον, ε, με το σχέδιο προπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν ε, οι δαπάνε του 2015 και κυρίω να αντιμετωπιστεί και η κρίση από το ρωσικό εμπάργο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα και ένα γεγονό που θα πρέπει να το έχουμε συνεχώ κατά νου. Δεύτερο βασικό συμπέρασμα. Η διορθωτική επιστολή αφορά την επαλληλία της χρηματοδότησης για τα έκτακτα μέτρα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες αναδιάταξης που έχουμε και να χρησιμοποιήσουμε το αποθεματικό πρόβλεπτο των αναγκών ως έσχατο μέσο, μόνο εφόσον χρειαστεί και για τα συγκεκριμένα ποσά. Επίσης, να διαφυλάξουμε το διαθέσιμο περιθώριο στο Γεωργικό Ταμείο και το δεύτερο, το δεύτερο ανατοτόριο για μελλοντικές κρίσεις. Επίσης, ε, το θέμα της ε, ε, παρουσίας της κρίσης στο δεύτερο εξάμεινο. Για τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε κάποια χρήματα στην άκρη ή σε περίπτωση που δημιουργηθούν έκτακτες ανάγκες ή επιτακτικές ανάγκες σε άλλα τμήματα του προπολογισμού να μπορούμε να κάνουμε ανακατανομές. Προτείνουμε λοιπόν ανακατανομή κάποιων πιστώσεων πληρωμών για να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες αλλού, ιδιαίτερα ε, για να καλυφθούν ανεξάφλητοι λογαριασμοί στα προγράμματα 1α, ε, του τομέα 1α, του τομέα 2 και του τομέα 4. Ευχαριστώ και με στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε απορίες σας. Σας ευχαριστώ κυρία μου για την ανάπτυξη του θέματος. Πράγματι τεχνικό θέμα. Το σχέδιο, το σχέδιο διορθωτικής επιστολής προκαλεί κάποια ερωτηματικά ανησυχίες αλλά και διαμαρτυρίες. Θα χρειαστεί λοιπόν να προσαρμόσουμε την τεχνική επιχειρηματολογία στον πολιτικό λόγο. Και αυτό είναι και το νόημα της σημερινής συνταλλαγής απόψεων. Και τώρα έχουμε και, τους, ε, μάλλον έχουμε και την παρουσία των μελών της Επιτροπής Γεωργίας. Η κυρία Γιάχτεν Μάκη έχει ζητήσει το λόγο. Έχει το λόγο, κυρία. Παρακαλούμε το μικρόφωνο. Θα μιλήσω φιλανδικά. Γιατί είναι πράγματι τεχνική η ορολογία του θέματος και θα μιλήσω λοιπόν στην μήτρική μου. δεν θα μπορούσα να εκφραστώ σε άλλη γλώσσα, στα γαλλικά τουλάχιστον δεν θα μπορούσα και ιδίω μιας και είμαι νέα ευρωβουλευτή. Ίσως να μην μπορέσω να χρησιμοποιήσω τους σωστούς τεχνικούς όρους, ελπίζω όμως ότι το μήνυμα θα περάσει. Με απασχολεί ιδιαίτερα η κρίση που προκαλούν οι ρωσικές κυρώσεις. Πώς θα αντισταθμίσετε την ζημία των γαλακτοπαραγωγών. Πώς θα αποζημιωθούν για τη ζημία που υφίστανται και πότε. Το Συμβούλιο Γεωργίας και ο προηγούμενος Επίτροπος είπαν ότι η γαλακτοπαραγωγή των βαλτικών χωρών και της Φιλανδίας θα έπρεπε ήδη να είχαν λάβει αποζημίωση, πακέτο αποζημίωσης από φέτος. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει άλλα πράγματα και βλέπω να προτείνει μεταφορές πιστώσεων για την καταπολέμηση του ιού έμπολα και άλλα σχετικά. Πολύ σημαντικά βέβαια θέματα, δεν αμφιβάλλω, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση α, υποσχέθηκε να αποζημιώσει τους γαλακτοπαραγωγούς. Θα πρέπει λοιπόν να τηρήσει τα υπεσχημένα. Και η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί φέτος. Άκουσα με ικανοποίηση ότι το πακέτο της αποζημίωσης μάλιστα φαίνεται να διαμορφώνεται και υπερβολικά γενναιόδωρο. Τόσο το καλύτερο. Αλλά γιατί τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει την απόφαση αυτή και αφαιρεί χρήματα από το πακέτο αποζημιώσεων για να τα διαθέσει αλλού. Οι αγρότες βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση. Άλλοι έχουν αποζημιωθεί, άλλοι όχι. Οι νότιοι δρούν ταχύτερα. Αλλά δεν μπορεί να είναι σωστό αυτό. Όταν έχουν δοθεί υποσχέσει, αυτές πρέπει να υλοποιηθούν. Γι' αυτό και ρωτώ, γιατί γίνονται οι μεταφορές αυτές πιστώσεων. Ελπίζω ότι θα καταβληθούν οι αποζημιώσει το ταχύτερο δυνατό, διότι οι ζημίες είναι πολύ μεγάλες. Θα οδηγηθούν και σε πτωχεύσει σε ορισμένες και είναι εν τέλει και ζήτημα αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο θα πιστέψει τι υποσχέσει τη πλέον. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γυριάντα. Σας ευχαριστώ. Εμεί, οι Ιρλανδοί δηλαδή, έχουμε σημαντικές επιφυλάξεις. Το ποσό της κρίσης θα ληφθεί από άμεσες πληρωμές. Και τα, μέσα τα μέτρα για τη Ρωσία μας αφήνουν μοναχά... Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετά τώρα ειδικό πακέτο αποζημιώσεων για τους γαλακτοπαραγωγούς της Φιλανδίας και των Βαλτικών χωρών. Θα έχει τεράστια όμως επίπτωση αυτό στην Ιρλανδία που είναι βεβαίως αγροτική η οικονομία της. Και τελικά οι αγρότες μας θα αντιμετωπίσουν προβλήματα από τη μείωση του 1,3%. Ήδη έχουμε κρίση με το βόλιο κρέα στην Ιρλανδία. Έχουμε ούτω ή άλλω και κρίση τη αγροτική οικονομία και των τιμών που πέφτουν δηλαδή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανησυχούμε λοιπόν ότι οποιασδήποτε περαιτέρω περικοπέ από το Γεωργικό Ταμείο. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ο προπολογισμό αντιμετωπίζει σοβαρέ πιέσει σε, όλες, σε όλους τους τίτλους του, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε πώς είναι δυνατόν να αφαιρεθούν χρήματα από το Γεωργικό Ταμείο για να δοθούν αλλού. Δεν είναι λύση αυτή. Τρίτη ερώτηση και μετά ας απαντήσει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξηγήσει ε, που μας έδωσε και να πω ότι η ζήτηση αυτή είναι κέρια σημασία για να αποφασίσουμε έχοντας γνώση της κατάστασης. Η πρώτη μου ερώτηση είναι καθαρή και εξάστερη. Έχουμε άμεσα κάποιες ε, ζημίες για τους γεωργούς από τη συγκεκριμένη διορθωτική επιστολή. Θα πλήξει συγκεκριμένη επιστολή διορθωτική τους γεωργούς. Και το 2015, σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κρίση, υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να επιτρέπει την αποζημίωση των ε, γεωργών είτε εξαιτία του ρωσικού εμπάργου είτε εξαιτία άλλη κρίσης. Ερωτώ λοιπόν συγκεκριμένα, τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που δεν, δεν επαρκέσει το αποθεματικό των απρόβλεπτων αναγκών της κρίσης για να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις. Τι προτάσεις έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς ε, θα μας ε, καθησυχάσει ότι από αυτή τη διορθωτική επιστολή θα προκύψουν ούτε άμεσες ζημίες, ούτε μεταγενέστερες ζημίες για τους γεωργούς. Και επαναλαμβάνω, αν συνεχιστεί το ρωσικό εμπάργο ή αν ανακύψει νέα κρίση, τι θα γίνει, τι μέτρα θα αναλάβει η Επιτροπή σε περίπτωση που κρυθούν ανεπαρκή τα κονδύλια της κρίσης απρόβλεπτων αναγκών. Ευχαριστώ. Θα πρότεινα να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Καλβίνια για να απαντήσει και μετά θα συνεχιστούν οι ερωταπαντήσεις. Κύριε Καλβίνιο, παρακαλώ. Προσέξτε το ρυθμό σας. Slow, παρακαλώ. Yes, thank you very much. Thank you very much. Ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφου σας για τις ερωτήσεις που όντως απηχούν τις αντιδράσεις που έχουμε ακούσει και εμείς και που είναι κατανοητές. Διότι όλο αυτό το engineering του προϋπολογισμού είναι πολύ περίπλοκο να εξηγηθεί. Αλλά πράγματι δεν ε, άπηχουν και την πραγματικότητα οι παρατηρήσεις αυτές του περιεχομένου δηλαδή της διορθωτικής επιστολής. Το πρώτο για τις αποζημιώσεις δηλαδή, των γαλακτοπαργογών. Να σας πω σαφώς ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει τίποτε ακόμα σχετικά με τον προϋπολογισμό 2014 για να μεταφέρει εισδήποτε πιστώσεις αλλού. Αυτό που συζητούμε είναι ο προϋπολογισμός του 2015 που είναι αυτός ο οποίος εκτελείται από τα μέσα Οκτωβρίου. Μιλούμε δηλαδή για τον προπολογισμό του επόμενου έτους. Δεν έχει γίνει καμιά ανακατανομή που να αφαιρέσει ποσά από τη Γεωργία. Στην ουσία ο προπολογισμό φέτος έχει και πλεόνασμα που θα μεταφερθεί βέβαια στο 2015 όπως σας είπα πριν. Οι αγρότες θα αποζημιωθούν. Όχι με τον παρόντα προπολογισμό, το φετινό δηλαδή, αλλά με τον προπολογισμό του χρόνου. Δεν έχει ληφθεί καμιά απόφαση που θα οδηγήσει σε καθυστέρηση της αποζημίωσης των Γιώργων και η διορθωτική επιστολή δεν έχει καμία επίπτωση σε οποιαδήποτε, δηλαδή ω επίπτωση οποιαδήποτε καθυστέρηση στην αποζημίωση των Γιώργων. Για το δεύτερο τώρα, όσον αφορά τις επιπτώσεις ε, πρόσθετων μέτρων στο αποθεματικό και εάν υπάρχει κάποιο ειδικό πακέτο για αποζημιώσεις. Όπως είπα πριν, πρέπει να εξετάσουμε την πραγματική, την, στην πράξη εφαρμογή δηλαδή των μέτρων. Τα μέτρα έχουν μεν εγκριθεί, βλέπουμε όμως μετά την εγκρισή τους ότι λόγω των περιστάσεων των αγορών οι αγρότες δεν έχουν ενδιαφερθεί, δεν τα βρήκαν ενδιαφέροντα τα μέτρα αυτά, δηλαδή δεν ε, επεζήτησαν την εφαρμογή τους. Όπως είπα πριν, σε ό,τι αφορά λοιπόν την εφαρμογή, 30% μονάχα των μέτρων για τα οποροκυπευτικά εφαρμόστηκαν. Και σταματούμε τα μέτρα για το γάλα, διότι δεν καταλήγουν σε εκείνους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, δηλαδή Βαλτικές χώρες και Φιλανδία. Γι' αυτό τώρα επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδικό πακέτο για να στοχεύσει μέτρα στο τομέα του γάλακτος για Βαλτικές χώρες και Φιλανδία. Αυτά βέβαια βρίσκονται στο στάδιο της προπαρασκευής και δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα απαντώ και στον κύριο Φερνάντες λέγοντας ότι η προσέγγιση μας είναι αυτή που βλέπετε στην διαφάνεια 9. Αν θέλετε μπορούμε να επανέλθουμε στη διαφάνεια 9. Να προβούμε σε μια διαδοχική εφαρμογή των χρηματοδοτήσεων για τα διάφορα μέτρα. Πρώτα να δούμε τις δυνατότητες ανακατανομής. Δεύτερο να χρησιμοποιήσουμε το αποθεματικό κρίσης μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και για τα ποσά όπου είναι αναγκαία. Τρίτο, έχουμε και ένα περιθώριο από το Γεωργικό Ταμείο Επιδοτήσεων για μελλοντικές κρίσεις. Αν δηλαδή τα ποσά τα οποία προβλέπουμε δεν είναι επαρκή και είναι αδύνατον να προβλέψει κανείς τι θα γίνει εάν η Ρωσία επεκτείνει τις κυρώσεις. Δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε όλα, τουλάχιστον όχι σε αυτή τη φάση. Παρ' όλα αυτά έχουμε ένα διαθέσιμο περιθώριο το οποίο μπορεί να κινητοποιηθεί με έναν τροποποιητικό προπολογισμό. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το τίτλο, έχουμε και τι περισσότερε εγγυήσει για να αντιμετωπίσουμε απρόβλεπτα γεγονότα και βεβαίω απόλυτα δικαιολογημένα. Έχουμε τι πιστώσει του προπολογισμού, έχουμε το περιθώριο, το οποίο θα μείνει κάτω από την ανώτατη οροφή του ε, Γεωργικού Ταμείου, έχουμε και άλλους μηχανισμούς που έχουν ως στόχο να, βοηθήσουν στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων το 2014. Αλλά δεν θα προσφύγουμε στο αποθεματικό της κρίσης αν υπάρξουν άλλα διαθέσιμα μέσα πριν. Θα ακολουθήσουμε μια διαδοχική σειρά εφαρμογών των μέτρων μέχρι ότου δούμε ποιο είναι το καταλληλότερο. Για να απαντήσω την τελευταία ερώτηση τώρα. Εάν η κρίση συνεχιστεί και ο προπολογισμό όπως τροποποιηθεί τώρα με την διορθωτική επιστολή δεν είναι επαρκής, θα έχουμε ακόμη ένα περιθώριο κάτω από την οροφή που θα προτείνουμε με ε, σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού να κινητοποιηθεί για του χρόνου βεβαίω. Ξανά αρχίζουμε τις ερωτήσεις. Κύριε Ντονανό, έχει χυθεί πολύ μελάνη για την διορθωτική επιστολή και έχει απασχολήσει πολύ και τον ειδικό τύπο της Γεωργίας. Η δημοσιονομικοί μηχανισμοί είναι βέβαια περίπλοκοι, το είδαμε και σήμερα, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι να διατηρήσουμε την αγροτική οικονομία, την γεωργία στην Ευρώπη. Θα δούμε εάν θα συνεχιστεί η κρίση αυτή από τις ρωσικές κυρώσεις και το 2015. Παραμένουν πολλές αβεβαιότητες ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να τηρήσει τα υπεσχημένα κυρίω μέσα στα πλαίσια της κοινή αγροτική πολιτικής, διότι πρόκειται εν τέλει για την ίδια την αξιοπιστία της. Εάν κινητοποιήσουμε από πριν το αποθεματικό κρίση είναι αλήθεια, ότι διατρέχουμε τον κίνδυνο, διατρέχουμε κινδύνους για το μέλλον, διότι ελοχεύουν και άλλες κρίσεις. Και στη Γεωργία και για το γάλα ιδιαίτερα και για τα απορροκυπευτικά, όπω μπορώ να πω εγώ για τη δική μου εκλογική περιφέρεια, η, το άνοιγμα της αγοράς της μολδαβία κινδυνεύει να οδηγήσει σε ανατροπή ισορροπιών για το θέμα του κρέατος, για το θέμα του γάλακτος, με το τέλος των ποσοστώσεων του γάλακτος και με το άνοιγμα του ανταγωνισμού βεβαίως, κινδυνεύουμε να δούμε και μια πλεονασματική παραγωγή που ενδέχεται να οδηγήσει την Ευρώπη σε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Εγώ τα έχω πει αυτά εδώ και μια πενταετία εδώ. Η κρίση του γάλακτος μπορεί να έχει και μια απρόσμενη επίπτωση στο βόλιο κρέας. Διότι το βόλιο κρέας συχνά είναι υποπροϊόν της γαλακτοπαραγωγής. Θα μπούμε λοιπόν τώρα σε πλήρη ανταγωνισμό με άλλους παραγωγούς και εμένα με ανησυχεί πολύ το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας αν δεν μπορέσουμε να προβλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις οι οποίες είναι δυνατόν να προβλεφθούν από τώρα. Τώρα να κινητοποιήσουμε ολόκληρο το αποθεματικό κρίσος για να αντιμετωπίσουμε ε, το πρόβλημα σήμερα, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν υπεύθυνο εκ μέρους μας. Μόλις έλαβα ένα μήνυμα από την κυρία Καρτιασάμπαλ που εξαιτία τη καθυστέρηση τη δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση. Πάντως, μα παρακαλεί να μην λάβουμε σήμερα απόφαση για την διορθωτική επιστολή και να αναβάλουμε τη λήψη απόφασης ε, για την Πέμπτη το πρωί, τότε που θα προετοιμάσουμε και τη θέση μας για τη συνδιαλλαγή. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον το να βλέπουμε τα 484, 484 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία να είναι ένα εκτελεστικό μέτρο. Το θέμα είναι γιατί δεν το γνωρίζαμε κατά το παρελθόν αυτό. Προσπαθούμε να αποκομίσουμε περισσότερα χρήματα από το Συμβούλιο και τώρα τι συμβαίνει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν υπερβολικά ποσά στον προπολογισμό, κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε. Εδώ πρόκειται για τιμέ αγορά, πρόκειται για προσδοκίε. Αυτό όμω που παίζει ρόλο είναι ότι και ο προπολογισμό το του 2015 ε, θα έχει τα ίδια ε, πλασματικά ποσά όπως και το 2014. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να ρωτήσω. Το δεύτερο αφορά στη βοήθεια λόγω του ρωσικού εμπάργου. Είπατε προηγουμένως ότι η Κομισιόν αυτή την ε, ενίσχυση μάλλον έχει αναχαιτήσει, έχει έρει κάποιες αιτήσει ε, επειδή υπάρχουν ε, κάποιες υποψίες απάτης, όχι μόνο στο τυρί, αλλά και σε άλλα προϊόντα. Και γνωρίζουμε ότι ορισμένες χώρες για μεμονωμένα γεωργικά προϊόντα έχουν ζητήσει περισσότερες ενισχύσεις από ότι κατ' ουσίαν θα δικαιούνται λόγω της συνολικής παραγωγής στη χώρα τους. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω γιατί η Κομισιόν συνεχίζει να καταβάλει αυτές τις ενισχύσεις παρότι υπάρχουν υποψίες για απάτη. Και το ότι λέγεται ε, ναι στο τέλος του χρόνου λόγω των διορθωτικών ποσών θα ε, διεκδικήσουμε πίσω τα χρήματα, αυτό δεν είναι μια ικανοποιητική απάντηση. Γιατί ξέρετε, εμάς δεν μας είναι αδιάφορο το κατά πόσον οι φορολογούμενοι πρέπει να καταβάλουν κάποια ποσά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβεί σε απάτες και μιλάμε επίσης ε, για ποσά τα οποία είτε είναι στον αθηνικό προπολογισμό είτε στον κοινωνικό προπολογισμό επιβαρύνουν όλους τους προλογούμενους. Γι' αυτό δεν μας είναι αδιάφορο το θέμα. Εγώ στις συζητήσεις που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έλεγαν κοιτάξτε ε, μην ανησυχείτε ε, θα σας δώσουμε πίσω τα χρήματα αν υπάρχει απάτη. Το θέμα όμω είναι ότι υπάρχουν αυτές οι υποψίες απάτης και τα κράτη-μέλη να το ξέρουν αλλά να κλείνουν τα μάτια. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε πάρα αυτά και αυτές είναι δύο ερωτήσεις τις οποίες είχα να υποβάλω. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ντες που είναι μέλος τη Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, είμαι 10 χρόνια ευρωβουλευτή. Ε, για πρώτη φορά είμαι μέλο τη Επιτροπή ε, Προπολογισμών και για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβω το πλαίσιο. Και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν παρήσατε στην συνάδελφο μου Πιντεγιά, ο οποίο ασχολείται με θέματα προπολογισμού στην Επιτροπή Γεωργία. Θα ήθελα όμω να επισημάνω κάποια θέματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Κομισιόν χρειάζεται τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να βοηθήσει του γαλακτοπαργωγού ε, στη Φινλανδία και σε άλλε σκανδιναβικέ χώρες. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές δεν κατανοεί κανείς όλες αυτές τις περίπλοκες διαδικασίες. Μίλησα για, με τον Φινλανδό και με τον Λονό Υπουργό Γεωργίας ε, και νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα πιο κατανοητό σύστημα αντισταθμίσεων. Ε, πριν από την κρίση ε, ήξερα και μίλησα για την τιμή γάλακτος στη Λετωνία, στη Φινλανδία και αμέσως μετά το μποϊκοτάρισμα λόγω των εξολήξεων στη Ρωσία είχε αλλάξει δραματικά η τιμή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε δύο μήνες μειώθηκε ριζικά αυτή η τιμή του γάλακτος, απειλείται η επιβίωσή τους και δεν ξέρω ποια είναι η λύση που μπορεί να προσφερθεί σε αυτού του αγρότες. Εγώ πρώτη ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα. Η κυρία Κρέσλε λέει ότι πρέπει να έχουμε υποψίες απάτη. 14 ήταν, 20 ήταν και τώρα 14, άρα 6 σέντη διαφορά ε, σε όλους, για όλου του ε, ε, για γαλακτοπαραγωγούς μειώθηκε η τιμή. Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξουν επιστροφές σε αυτή τη χώρα. Δίδεται όμως μόνο το 50%. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να κάνουμε όλου αυτού του υπολογισμού. Από ό,τι φαίνεται όμω στην Ευρώπη χρειαζόμαστε χρόνο. Ακριβώ αυτού, του ε, γεωργού τη Βαλτική, πρέπει να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα λόγω τη κρίση με τη Ρωσία. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσουμε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν το καταφέρνουμε. Και οι συγκεκριμένοι γεωργοί θα καταστραφούν αν δεν λάβουν ενισχύσει αμέσω επόμενε εβδομάδε. Ε, από τη δική μου τη χώρα, την Βαβαρία, επίση ε, διεκδικούμε ενισχύσεις. Ε, βέβαια, εγώ δεν είμαι εκείνο που λέω πάντα θα πρέπει να πληρώσει ο φορολογούμενος. Όπου όμως υπάρχουν προβλήματα για την επιβίωση και υπάρχουν πολιτικά αίτια λόγω αυτού, τότε θα πρέπει να δραστηριοποιείται η Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση στον προπολογισμό, αποκινούμε τον κύριο Ντεκάστρο από τους ε, σοσιαλιστές ε, αλλά και με άλλους ε, συναδέλφους απέστειλα μια επιστολή προς τον πρόεδρο κύριο Γιούγκερ και λέω ότι δεν είναι δυνατόν κονδύλια τα οποία έρχονται πίσω στον προπλογισμό να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. 400 εκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο της Κρίσης. Τι είναι αυτό. Αυτό δεν είναι τίποτα όταν υπάρχει πραγματική κρίση. Έχει κάνει κανείς υπολογισμούς πώς ακριβώς θίγονται οι γαλακτοπαραγωγοί στην Ευρώπη όταν μειώνεται τόσο δραστικά η τιμή. Μιλάμε για 5,6 δις ευρώ και όταν μιλάμε για ακόμα ριζικότερη μείωση ε, το ποσό είναι ακόμα μεγαλύτερο. Άρα δηλαδή αυτά τα ελάχιστα ποσά τα οποία προβλέπονται δεν μπορούν να βοηθήσουν. Εγώ δεν είμαι βέβαια εμπειρογνώμονας, αλλά δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο να αυξάνονται τα ποσά, να μην γίνεται η τελική αποζημίωση και η καταβολή στο τέλος του έτους και κάποια στιγμή δεν θα έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια για την αντιμετώπιση της κρίσης. Εγώ λοιπόν τάσομαι υπέρ του ότι τα κονδύλια τα οποία προβλέπονται για τον γεωργικό τομέα να παραμείνουν σε αυτό το γεωργικό τομέα και να διατεθούν στους γαλακτοπαραγωγούς στις χώρες της Βαλτικής και στη Φιλανδία. Ακριβώς γιατί και αυτοί πρέπει να πιστεύουν στο μέλλον της Ευρώπης. Κύριε Καλεβίνιο. ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με τις πολιτικές δηλώσεις ε, για την ανάγκη να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, τις υποσχέσεις μας, να προσπίσουμε την κοινή πολιτική. Επί της αρχής δεν διαφωνούμε καθόλου. Το θέμα είναι πώς θα υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους με το ελάχιστο δυνατό κόστος δεδομένων των δημοσιονομικών μας περιορισμών και των αντίξεων δημοσιονομικών συνθήκων. Κύριε Γκρέσλε, Έχω δύο παρατηρήσεις. Το γεγονός ότι υπάρχει πλεόνασμα στον γεωργικό προϋπολογισμό δεν μας εκπλήσει. Γιατί δεδομένου ότι έχουμε όλα αυτά τα μέσα και τους μηχανισμούς που θα πληρωθούν στα τέλη του έτους, είναι λογικό που κάθε χρόνο καταλήγουμε, ολοκληρώνουμε το δημοσιονομικό έτος με πλεόνασμα. Έχουμε γύρω στα 900 εκατομμύρια φέτος πλεόνασμα. Ένα τμήμα του αφορά την, ε, ε, επιστρο... τις επιστροφές από τη δημοσιονομική πειθαρχία ή το χρησιμοποιεί το αποθεματικό της κρίσης. Είναι φυσιολογικό λοιπόν που στα τέλη του έτους έχουμε ένα πλεόνασμα που είτε θα επιστραφεί είτε θα μετακυληθεί στον επόμενο προϋπολογισμό ανάλογα με τις συνθήκες. Στόχος μας είναι να προβλέψουμε τα έσοδα ειδικού προϋπολογισμού για το 2015 χάρη στις διορθώσεις που θα γίνουν για τις δαπάνες. Οι διορθώσεις λοιπόν που είναι δημοσιονομικές διορθώσεις και είναι αντικείμενο συζήτηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών θα οδηγήσουν σε αυξημένα έσοδα ειδικού προορισμού του χρόνου. Και δεν έχει νόημα να ολοκληρώσουμε το 2015 με επιπλέον πλεόνασμα ακριβώς επειδή θα έχουμε χρησιμοποιήσει επαρκώς αυτά τα ειδικά, έξοδα, τα ειδικά έσοδα στη διάρκεια του έτους. Σε ό,τι αφορά τις υπόνοιες απάτης, εγώ δεν έχω καμία πληροφορία που να υπενήσετε τέτοιες υπόνοιες απάτης. Μερικά μέτρα δεν ήταν επαρκώς στοχοθετημένα, ήταν υπερβολικά γενικά και ίσως α, και κάποιους γιοργούς που δεν τα κατανάγει εξαγωγής προς τη Ρωσία. Δεν, ε, δεν ήταν απάτη λοιπόν με στην έννοια. Απλώς το μέτρο ήταν υπερβολικά γενικό, δεν ήταν αρκετά στοχοθετημένο και προσανατολισμένο και έτσι υποφελήθηκαν και μερικοί που ίσως ε, δεν θα έπρεπε να υποφεληθούν. Με ρωτήσατε γιατί δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη τα μέτρα για τη Φιλανδία και τις βαλτικές χώρες. Δεν οφείλεται κάτι τέτοιο στην αργοπορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γίνονται σφοδρές συζητήσεις ε, συνεχώς στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Θέλουμε όμως αυτά τα μέτρα να είναι σωστά στοχοθετημένα και γι' αυτό χρειαζόμαστε αντικειμενικά κριτήρια που θα προβλέπουν τους επιλέξιμους γεωργούς που θα επωφεληθούν από τα μέτρα αυτά. Και μερικά ζητήματα είναι αρκετά περίπλοκα. Για παράδειγμα, ένας από τους δείκτες είναι η αντικειμενική τιμή. Η αντικειμενική τομή όμως ε, στην ε, τιμή στην φιλανδική αγορά είναι σχετικά υψηλή. Οπότε δεν έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που να δικαιολογεί τη λήψη μέτρων. Τέτοιου είδου θέματα εξετάζονται αυτή τη στιγμή από του Υπουργού Γεωργία. Γι' αυτό και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη το σχετικό πακέτο, δεν έχει εγκριθεί το πακέτο βοήθεια προ τη Φιλανδία και τι Βαλτικέ χώρε. Παρόλο που υπάρχει πολιτική βούληση να βρεθεί μια σωστή, δίκαιη και στοχοθετημένη λύση για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου αυτού προβλήματο. Ευχαριστώ. Merci, ευχαριστώ. Ο κύριος Κούσμουκ. Ευχαριστώ. Βέβαια η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Είχαμε τις ρωσικές κυρώσεις, το ρωσικό εμπάργο που εξακολουθεί να ισχύει ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να μεταφερθεί το αποθεματικό κρίσης στο επόμενο έτος παρόλο που ίσως θα ήταν η μόνη δυνατότητα που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις ζημίες από το ρωσικό εμπάργο. Νομίζω ότι στηρίζεται σε μια μεγάλη παρεξήγηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί οι συνέπειες της, των ρωσικών κυρώσεων είναι η σημαντική μείωση των τιμών. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, είχαμε σημαντική μείωση. Μερικές φορές 30-40%, ε, μερικές φορές μέχρι και 70% είναι η μείωση των τιμών σε σχέση με τις τιμές που είχαμε πριν από την κρίση και το ρωσικό εμπάργο, τις ρωσικές κυρώσεις. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι τα φετινά κονδύλια για τις αποζημιώσεις δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο έπακρο, ενώ η οι αποζημιώσεις που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ενισχύσεις που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είχαν ακριβώς τέτοια διάρθρωση ώστε οι αποζημιώσεις να ωφελήσουν πολύ λίγους γεωργούς. Σε ό,τι αφορά τα απορροκυπευτικά, οι αποζημιώσεις αυτές ε, ε, υποβλήθηκαν, δόθηκαν είτε σε γεωργούς που μειώνουν τις, τις καλλιέργειές τους, είτε που δίνουν τα απορροκυπευτικά τους για φιλαθροπικό σκοπό. Και είναι ε, λίγοι γεωργία αυτή, Ενώ κανονικά τα μέτρα θα πρέπει να ωφελούν όλους τους γεωργούς ε, που εξήγαγαν προς τη Ρωσία και όχι ένα μικρό τμήμα τους μόνο. Και επισημαίνω ότι το, το πρόβλημα αυτό δεν ε, αφορά μόνο τη Φιλανδία και τις βαλτικές χώρες. Οι Πολωνοί γεωργοί είχαν ε, ο γύρω γύρω στα 500 εκατομμύρια ε, από τις εξαγωγές προς τη Ρωσία. Οπότε το ρωσικό εμπάργο έπληξε ε, και τους Πολωνούς Γεωργούς και μάλιστα πολύ σοβαρά. Θα ήθελα λοιπόν να αποτρέψω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το να μεταφέρει το αποθεματικό της κρίσης στον επόμενο έτος. Νομίζω ότι είναι μεγάλη παρεξήγηση το όλο σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην χρησιμοποιήσει το έπακρο φέτος το αποθεματικό κρίσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις και να δώσει κάποιες εξηγήσεις η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούσαμε ότι ήδη δόθηκαν αποζημιώσεις για το ρωσικό εμπάργο, ενώ άλλες αποζημιώσεις δεν έχουν ακόμη καταβληθεί. Γιατί ε, εκκρεμούν ακόμη αποζημιώσεις που θα πρέπει να χορηγηθούν για να διορθωθούν ε, οι ζημίες από τις ε, ρωσικές κυρώσεις. Και αν δεν έχουν εκταμιευθεί οι σχετικές αποζημιώσεις, γιατί αυτή η καθυστέρηση, πού οφείλεται αυτό. Γιατί και εμείς στην ε, Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν γνωρίζουμε αν έχουν καταβληθεί όλες οι αποζημιώσεις οφειλόμενος ή ή όχι γιατί προκύπτει ότι δεν έχουν καταβληθεί ακόμη όλες οι αποζημιώσεις. Επίσης υπάρχει και θέμα ορισμού. Για μας στην Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι σημαντικό να ορίσουμε πολύ αυστηρά τι εστί αποθεματικό κρίσης. Γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει αποθεματικό κρίσης. Το ρωσικό εμπάργο, οι ρωσικές κυρώσεις δημιούργησαν κρίση στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική. Γιατί αν όντω δημιούργησαν κρίση, τότε θα πρέπει να κινητοποιήσουμε το αποθεματικό της κρίσης. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει κρίση και άρα θα πρέπει να κινητοποιήσουμε αυτό το αποθεματικό. Το θέμα είναι για ποιο ποσό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι για το χρόνο θα χρειαστούν 350 εκατομμύρια για το αποθεματικό αυτό. Πώς κατέληξε σε αυτόν τον υπολογισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν α, ε, κατάλαβα ακριβώς ε, πώς προέκυψε αυτός ο προϋπολογισμός. Νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα με τον ορισμό της έννοιας του αποθεματικού της κρίσης. Γιατί κατά τη γνώμη υπάρχει κρίση και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτό το αποθεματικό. Τώρα σε τι ποσό αυτό είναι θέμα ανάλυσης. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους που παρακολουθούν το έργο μας να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Είπαμε ότι το αποθεματικό της κρίσης σε ύψος 1% προκύπτει από τις άμεσες ενισχύσεις. Οι συνάδελφοι όμως και είπαν ότι οι ίδιοι οι γεωργοί θα πληρώσουν τα σπασμένα της κρίσης και των κυρώσεων. Ήδη θα πρέπει να το χρηματοδοτήσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι ό,τι θα πληρωθεί από το αποθεματικό της κρίσης κατά τα τέλη του 2015 θα επιστραφεί στους γεωργούς με το προβλεπόμενο πλεόνασμα που αναμένουμε για τα τέλη του έτους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το καταλάβουν οι γεωργοί. Θα πρέπει να εξηγήσουμε αν αυτό το πλεόνασμα θα τους αφαιρεθεί θα αφαιρεθεί από τις άμεσες ενισχύσεις και μετά προς το τέλος του έτους θα επιστραφεί και μάλιστα με το, υπερ, με το πλεόνασμα. Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσεις για όλα αυτά τα θέματα. Αν έχουν καταβληθεί όλες οι αποζημιώσεις ή όχι. Ορισμός του αποθεματικού της κρίσης. Και τα χρήματα που θα αφαιρεθούν από το αποθεματικό της κρίσης θα επιστραφούν κάποια στιγμή στους ε, γεωργούς και μάλιστα με τα πλεονάσματα. Αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόλμελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά αυτό το σχέδιο για το οποίο συζητάμε σήμερα, εμένα μου προκάλεσε έκπληξη με την εξή έννοια, ότι εμφανίστηκαν κάποια κονδύλια τα οποία υπάρχουν στη διάθεσή μας, τώρα όμως καταλήγω στο ότι τελικά ε, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς ε, τι συζητάμε γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αστάθμητοι παράγοντες και διάφορες συγκεχημένες απόψεις ε, που κατά κάποιον τρόπο βέβαια αυτοί που τις προβάλλουν προσπαθούν να τις αιτιολογήσουν. Και η εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι αυτή είναι μια πεπατημένη, μια συνήθιση διαδικασία. Πρέπει όμως να σας πω ότι εγώ αν τα πράγματα είναι έτσι τότε δεν καταλαβαίνω γιατί στην Επιτροπή τίθενται τόσα πολλά ερωτήματα. Πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η διαδικασία για την υποτίθεται συνηθισμένη ε, συζήτηση που γίνεται. Και θέλω να σας πω το εξής. Νομίζω ότι πρέπει να είναι σε όλους μας σαφές ότι χρειαζόμαστε ένα διαφανή προϋπολογισμό που σημαίνει ότι μπορούμε να προβούμε σε εκταμείευση κονδυλίων μόνο εφόσον η κατάσταση είναι σαφής. Αυτό για μένα σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια βάση υπολογισμού. Αυτή τη στιγμή ακούμε να εκτοξεύονται διάφορα ποσά ας πούμε, για διάφορους ε, τομείς ε, δαπανών, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια σωστή βάση υπολογισμού για την εκταμείευση πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αξιοπιστία. Δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος ε, δικαιούται να ισχυρίζεται ότι υπολογίζει στις υποσχέσεις μας, ε, πρέπει και να δικαιώνεται. Πρέπει οι υποσχέσεις να τηρούνται. Εκτός αυτού, μιλάμε για αποθεματικό και βλέπουμε ότι έρχονται και επανέρχονται οι κρίσεις, ε, όπως παραδείγματος χάνει τώρα στο θέμα των μέτρων κατά της Ρωσίας και είναι αυτονόητο ότι και εγώ πιστεύω ότι πρέπει κανείς ε, να βοηθήσει αμελητή τους άμεσα θυγόμενους. Αλλά για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε στον προπολογισμό αποθεματικά. Αλλιώς δεν θα μπορούμε να βοηθήσουμε στον δεχόμενο των μελλοντικών κρίσεων. Άρα δηλαδή καταρχήν χρειαζόμαστε ένα σαφώς δομημένο πακέτο το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει εναλλακτικέ λύσεις οι οποίες βέβαια και αυτές με τη σειρά τους πρέπει να είναι σαφείς για να μπορούμε να ψηφίσουμε αλλά σας είπα στο πλαίσιο ενός συνολικού πακέτου. Κυρία Καλβίνια, θέλετε να απαντήσετε στη σωρία ρωτήσω που υπέβαλαν οι συνάδελφοι. Yes. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι Καταρχήν, θέλω να σας πω το εξή ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ευρωβουλευτή που ισχυρίστηκε ότι η κρίση έπληξε κυρίως την Πολωνία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η Πολωνία υποφελήθηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος από την πρώτη δέσμη μέτρων για τα οποροκυπευτικά. Μιλάμε για περίπου το 40% αυτών των μέτρων που διοχετεύτηκαν στην Πολωνία και γι' αυτό χρειαστήκαμε ένα δεύτερο πακέτο για να καλύψουμε τις ανάγκες των υπόλοιπων μελών. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει σαφή συσχετισμό ανάμεσα στι χώρε που επλήγησαν περισσότερο και στα μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν. Όσον αφορά τώρα το κατά πόσον υπήρξε εξόφληση των, ε, των κρεμουσών πληρωμών, θέλω να σας πω ότι ο Ευρωπαϊκός Προπλογισμός προβλέπει την αποζημίωση των κρατών μελών μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που είναι κατά κανόνα γύρω στους δύο μήνες. Έχουμε λοιπόν ένα πρώτο, μια πρώτη δέσμη μέτρων που προβλέπει κάποιες αποζημιώσεις. Αυτές θα ολοκληρωθούν νομίζω σύντομα. Θα δω ποιες είναι ακριβείς ημερομηνίες. Εν περιπτώσει τώρα φτάνουμε στην στιγμή επιστροφής κονδυλίων προς τα κράτη-μέλη και το δεύτερο πακέτο εξακολουθεί να τρέχει. Άρα δηλαδή αυτή στιγμή τα κράτη-μέλη καταβάλουν τα ποσά τα οποία μετά θα επιστραφούν από τον ε, ενωσιακό προϋπολογισμό. Το τρίτο ερώτημα αφορά στο κατά πόσον αυτή η κατάσταση ε, καλύπτεται από το αποθεματικό της κρίσης. Βεβαίως και το αποθεματικό αυτό δεν χρηματοδοτήθηκε από τους γεωργούς γιατί και καμία κρίση δεν προκαλείται από τους γεωργούς. Άρα δηλαδή αυτό το αποθεματικό αφορά απρόβλεπτες εξελίξεις στην αγορά και κατά την άποψή μας και βεβαίως και από τις της Νομικής είναι ότι αυτό το σκηνικό υπάρχει τώρα, άρα δηλαδή το αποθεματικό της κρίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τώρα, κατά πόσον θα επιστραφούν τα ποσά του αποθεματικού στους γεωργούς ε, το 2015, αυτό είναι συνάρτηση των μέτρων που θα ληφθούν. Συνάρτηση επίσης ε, του κατά πόσον θα υπάρξουν κονδύλια για να εκταμιευτούν και θα εξαρτηθεί επίσης κατά πόσον θα έχουμε μεγαλύτερα ποσά ειδικού σκοπού για την επόμενη χρονιά από αυτά που προβλέπονται τώρα. Θα εξαρτηθεί επίσης, όταν θα φτάσουμε εκείνη τη χρονική στιγμή, από τους παράγοντες που θα επικρατούν, γιατί σήμερα δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα. Επίση δεν μπορούμε να προβλέψουμε το κατά πόσον θα εξαντληθεί πλήρω το αποθεματικό και δεν θα επιστραφεί καθόλου στους ε, αγρότε. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Όσον αφορά τώρα στη διαδικασία, για αυτή την ε, πεπατημένη όπω την αποκαλέσατε, χρειαζόμαστε πράγματι διαφάνεια ε, Κατά κανόνα αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή, γίνεται η επικαιροποίηση των εσόδων ειδικού σκοπού με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν των διορθώσεων της εισφοράς γάλακτος Άρα δηλαδή κατά κανόνα το φθινόπωρο εξετάζουμε αυτά τα στοιχεία, τα επικαιροποιούμε και κατόπιν υποβάλλουμε μια διορθωτική επιστολή. Αυτό όμω που έγινε ε, φέτο για πρώτη φορά και προκάλεσε τι αντιδράσει είναι, όπω σα είπα, για πρώτη φορά ε, αναφερθήκαμε στη δυνατότητα να γίνει χρήση του αποθεματικού κρίση και αντί να προστίθεται η μία, το ένα αποθεματικό πάνω στο άλλο και τα κονδύλια του προπολογισμού στα άλλα, αποφασίσαμε να εκταμιεύσουμε αυτά που αποφασίσαμε ότι δεν χρειαζόμαστε για την γεωρική πολιτική για άλλους τομείς του προϋπολογισμού. Για πρώτη φορά λοιπόν η δημοσιονομική πειθαρχία είναι εκείνη η οποία αρχίζει και, αρχίζει και να παρισφρεί στον τομέα της γεωργικής πολιτικής. Δεν μας εκπλήσουν βέβαια οι αντιδράσεις, αλλά επιθυμούμε να είναι σαφέ ότι ε, όσοι έχουν τώρα τα πράγματα στον προπολογισμό, δεν θα ήταν υπεύθυνο να αναδιατάξουμε τα υπάρχοντα κονδύλια για να γίνει η βέλτιστη χρήση των πιστώσεων πληρωμών που έχουμε στη διαδεσή μα και είναι πολύ λίγε. Επίσης, θέλω να πω ότι ναι, πράγματι χρειαζόμαστε αποθεματικό στον προπολογισμό κυρίως για τη γεωργική πολιτική. Το θέμα είναι το ύψος αυτού του αποθεματικού και εις βάρος ποιων άλλων τομέων ή ποιων άλλων στοιχείων του προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ. Θα ολοκληρώσουμε τώρα τον κατάλογο των αγορητών. Έχουμε τρεις ακόμη ομιλητές. Ο κύριος Μάνικα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλούμε για σημαντικά προβλήματα. Αυτό το δείχνουν και οι αντιδράσεις των συναδέλφων μου που εκφράζουν σημαντικές ανησυχίες και τις οποίες κατανοώ. Αν δεν συνδράμουμε τους αγρότες και για τις επιπτώσεις του εμπάργου των Ρώσων και, και που πρόκειται δηλαδή από τη σύγκρουση γύρω από την Ουκρανία θα δούμε σημαντικές παραμορφώσεις. Αυτό όμως που λείπει εδώ είναι μια συνολική εικόνα. Μιλήσαμε όμως τώρα για λογαριασμούς. Αν όμως δεν δούμε την εικόνα στο σύνολό της, το πρόβλημα θα παραμείνει και δεν θα λειτουργήσει η δομή που προσπαθούμε να φτιάξουμε. Συζητούμε τις επιπτώσεις των κυρώσεων. Τελικά όμως, πώς θα λυθούν τα προβλήματα με κρατικές επιδοτήσεις. Θα είναι η ίδια λύση σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν ε, οι τόκοι υπερημερίας που πρέπει να ρυθμιστούν και, αυτού, και αυτοί. Αυτά τα 25, μάλλον τα 2,5 δις, τον, τα 25, συγγνώμη, τα 25 δις του ελλείμματος που έχουμε μέχρι του χρόνου θα μας βασανίζουν ακόμη. Δεν ξέρω αν μπορεί να λυθούν αυτά μέσα σε τριμερή διάλογο. Ούτε από το Συμβούλιο, ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούω κάποιες προσεγγίσεις λύσεων. Κανείς δεν γνωρίζει τις πραγματικές επιπτώσεις της διορθωτικής επιστολής. Αυτή τη διορθωτική επιστολή λοιπόν πρέπει να τη δούμε μέσα σε αυτή τη συνολικότερη εικόνα. Σας ευχαριστώ κύριε Ταρών. Ευχαριστώ. Θα επαναλάβω κάποιες ερωτήσεις που ήδη τέθηκαν. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη... Είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα πριν από την συνδιαλλαγή. Βρισκόμαστε σε περιόδου κρίσεων, ιδίω στο γαλακτοκομικό τομέα. Και έχω μεγάλες αμφιβολίες αν πρέπει όντω να μειωθεί το αποθεματικό κρίσεως για τον επόμενο προπολογισμό. Και θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει άλλου τρόπου άμεσων χρηματοδοτήσεων για αποζημιώσει από το ε, ρωσικό εμπάργο. Η ομάδα μου κατανοεί βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει πολλές, ε, πολλούς περιορισμούς ε, δημοσιονομική πειθαρχία, λιτότητα και την οροφή του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ωστόσο έχω δύο απλές ερωτήσεις. Σωστά θεωρώ ότι το πρόσθετο εισόδημα του Ταμείου Εγγυήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πληρωμές στον προϋπολογισμό και όχι για υποχρώσεις και ότι συνεπώς το πρόσθετο αυτό εισόδημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο ρωσικό εμπάργο. Δεύτερο, πιστώσεις και υποχρώσεις μαζί μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς το αποθεματικό κρίσος. Τέλος, Μια και είμαι outsider για θέματα ε, αγροτικά. Η Κομισιόν έχει επικριθεί για την καθυστέρηση των αντιδράσεών της. Δύο μήνες έχουν περάσει ήδη. Για μας και βέβαια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο μήνες δεν είναι τίποτα. Τι να προλάβει να κάνει κανείς. Όμως για την Αγελάδα και για τον ιδιοκτήτη της Δύο μήνε είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Να το λάβετε υπόψη σα αυτό. Μάλιστα, σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κρίση της ε, Ρωσίας μας απασχολεί όλους γιατί ακούσαμε ότι υπήρξε τώρα μία συμφωνία με τον Επίτροπο Οτιγκερ έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει εγγυήσει για αγορές αερίου ε, στην Ουκρανία. Και με ενδιαφέρει πώς αυτό θα ληφθεί υπόψη στον προπολογισμό και κατά πόσον θα υπάρχουν αποθεματικά ε, και κατά πόσον ήδη δημιουργείται ένα αποθεματικό για αυτές τις πληρωμές. Κύριε Καλβινιό. Α, έχω. Κοιτάξτε, θα ήθελα να απαντήσω στις πολύ συγκεκριμένες και τεχνικές ερωτήσεις ε, που έθεσε Σιλβάνα σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Να εξηγήσω πώς αυτή λειτουργεί. Υπάρχει μια γενική εικόνα και πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα πρέπει να το εντάξουμε στην ευρύτερη εικόνα για τον προϋπολογισμό του 2015. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η γεωργία είναι ένας από τους τομείς όπου δεν υπάρχουν ανεξόφλητα ποσά. Δηλαδή, ε, κατά κανόνα κάτω από αυτό το πρίσμα εκεί δεν υπάρχουν εντάσεις. Και βεβαίως ε, εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι είναι εκείνο ο τομέας του προϋπολογισμού που μέχρι τώρα δεν είχε αντιμετωπίσει ένταση κάτω από αυτό το πρίσμα. Όσον αφορά τώρα τις αγορές αερίου στην Ουκρανία, πρέπει να πω στους συναδέλφους μου το εξή. Ε, και αν θέλετε μετά μπορούμε να το στήσουμε και σε διμερές επίπεδο. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, δεν το γνωρίζω. Ίσως ο, ο μπορεί όσον αφορά το θέμα, να σας πω το εξή. Τα έσοδα ειδικού σκοπού αφοράν, αφορούν πιστώσεις ε, πληρωμών ή πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Πρόκειται για δαπάνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο εγγύησεων για τη γεωργία δηλαδή και δεν είναι διαφοροποιημένες δαπάνες. Δηλαδή οι υποχρεώσεις και οι πληρωμές πηγαίνουν πάντα μαζί και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά τις εκταμιεύσεις για τον πρώτο πυλώνα της γεωργίας. Τα έσοδα ειδικού σκοπού θα μας υποχρεώσουν να έχουμε περισσότερες πιστώσεις πληρωμών και ανάληψης υποχρεώσεων. Η συνάδελφός μου σας εξήγησε ότι αν υπάρξουν περισσότερες επιστροφές ή εάν οι εφαρμογή του, των 45 δις ε, στο Ταμείο Εγγυήσεων για το 2015 αν αυτό το ποσό δεν χρησιμοποιηθεί πλήρως τότε θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πριν καταφύγουμε στο αποθεματικό κρίσης. Ας δούμε τώρα λιγάκι τη δημοσιονομική πεθαρχία. Υπάρχει. Καταρχήν υπάρχουν ε, οι πιστώσεις ε, στις, που έχουν προβλεφθεί στις συγκεκριμένες γραμμές του προεπλογισμού. Επίσης ε, μπορεί να υπάρξει κάποια υπέρβαση πάνω από αυτό που προβλέπεται τώρα στον, στη διορθωτική επιστολή. Κατόπιν υπάρχει η χρήση του αποθέματος κρίσης. Αυτή είναι η αλληλουχία των μέτρων και αν όλα αυτά δεν φτάσουν τότε θα καταρτιστεί και ένας διορθωτικός προϋπολογισμός ο οποίος ε, θα εκμεταλλευτεί τα κονδύλια που υπάρχουν κάτω από την οροφή του Γεωργικού Ταμείου. Έτσι θα διατεθούν τα επιπρόσθετα κονδύλια. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση και το σκηνικό που μπορούμε να προβλέψουμε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σαρβάμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ανακατανομής κάποιων κονδυλίων. Και τεχνικά τεχνικός πώς καταλαβαίνω το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη διορθωτική επιστολή. Αλλά από πολιτική άποψη θα πρέπει να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα γιατί ε, από πολιτική άποψη τα πράγματα είναι φως φανάρι. Τεχνικά είναι περίπλοκα αλλά πολιτικά είναι απλά. Νομίζω ότι θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα προς το Συμβούλιο ότι χρειάζεται ε, να επιδείξουν αλληλεγγύη τα κράτη-μέλη. Οι Γεωργοί δεν το ζήτησαν. Δεν ζήτησαν κάτι τέτοιο. Αλλά ως ε, υπήκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν τη συνένεσή τους ε, και είναι τμήματα της κοινή ε, πολιτικής, της κοινής γεωρικής πολιτικής. Αλλά όταν κατασταλάξουν τα πράγματα, όταν καταλαγιάσει ο κονιορτός, θα πρέπει να καθησυχαστούν οι γεωργοί και να φανεί αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό το μήνυμα θα πρέπει να στείλουμε στο Συμβούλιο. Αντιλαμβάνομαι το πολιτικό πρόβλημα. Τι τεχνικέ λεπτομέρειε θα πρέπει να τι αφήσουμε στου τεχνοκράτε. Και αυτό είναι το μήνυμα και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε στη μοίρα του τους Γιώργου. Παρόλο που από τεχνική άποψη είναι όλα άψογα και ω μέλο τη Επιτροπή Ιδιαλλαγή αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να πληρώσουμε του ανεξόφλητου λογαριασμού, αναφυσβήτητα, αλλά α μην ξεχνούμε το πολιτικό μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο ε, στον υποφαινόμενο να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις αν με επιτρέπετε. Αυτή η κατάσταση είναι η οδυνηρή ε, κατάσταση που δημιουργήθηκε από τους απλήρωτους λογαριασμούς. Αν δεν είχαμε τόσο, πολλού τόσο πολλούς ανεξόφλητους λογαριασμούς, δεν θα, είχε δεν ήταν αναγκαία η προσφυγή στη διορθωτική επιστολή εκ μέρου Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί εξαιτία από τον απλήρωτο λογαριασμό θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια ε, κονδύλια που προβλέπονταν για τη Γεωργία να τα ανακατανείμει αλλού. Και ναι, αν το πακέτο των διορθωτικών προπολογισμών για το 2014 περνούσε από συνδιαλλαγή και θα έπρεπε να το δεχτεί το αν το δεχόταν το Συμβούλιο αυτό το πακέτο, κυρία Καλβίνιο, θα είχατε αρκετά μέσα για να πληρώσετε τους λογαριασμούς. Σε ό,τι αφορά το αποθεματικό της κρίσης, πρόκειται για μια καινοτομία που συνδέεται με το ετήσιο το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο του 2014-2020. Για πρώτη φορά το 2014 συστήθηκε αυτό το αποθεματικό της κρίσης. Και αυτό το αποθεματικό κρίσης χρηματοδοτείται από την εισφορά των ε, δαπανών του πρώτου πυλώνα ε, από τα δικαιώματα παραγωγής. Ουσιαστικά οι ίδιοι οι γεωργοί χρηματοδοτούν αυτό το αποθεματικό της κρίσης. Είναι ένα σύστημα αυτασφάλισης ουσιαστικά που κάνουν οι γεωργοί. Οπότε η χρησιμοποίηση του αποθεματικού κρίσης για οποιοδήποτε άλλο στόχο που δεν αφορά τη γεωργία νομίζω ότι θα προκαλέσει εύλογες ε, επικρίσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Και μάλιστα διαγράφεται μια πολύ σοβαρή κρίση και στο γαλακτοκομικό τομέα και στον τομέα του κρέατος. Και οι προοπτικές τιμών είναι εξαιρετικά ανησυχητικέ. Και θα προκαλέσουν και στο εγγύς μέλλον ε, απρόβλεπτες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες. Οπότε θα πρέπει ήδη να προβλέψουμε κάποια αντισταθμιστικά μέτρα, κάποιες αποζημιώσεις για να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση πολλών γεωργών και κτηνοτρόφων. Αυτά και ο λόγος και πάλι στην κυρία Καλβίνιο για την τελευταία της παρέμβαση. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μας δώσατε για αυτή την ανταλλαγή απόψεων, που πραγματικά ήταν πολύ επικοδομητική και ενδιαφέρουσα. Γιατί πραγματικά έφερε στο επίκεντρο τα πιο σημαντικά θέματα, αυτά που αναφέρονται και στην διορθωτική επιστολή. Έχουμε επίγνωση του πολιτικού διακυβεύματος και σε καμία περίπτωση δεν διαφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί σας. Νομίζω ότι συνεργαζόμαστε για να βρούμε κατάλληλες λύσεις για τους Ευρωπαίους γεωργούς. Προτείνουμε λοιπόν κάποιες λύσεις, αλλά ταυτόχρονα είμαστε αρμόδιοι, επιφορτισμένοι με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Οπότε και στο μέλλον πιστεύω ότι όλο και περισσότερο ε, θα καλούμαστε να επιλύουμε τέτοια θέματα, γιατί φτάνουμε στον ε, σκληρό πυρήνα του προϋπολογισμού και θα έχουμε τέτοια προβλήματα στα πλαίσια του νέου πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Σας ευχαριστώ. Αυτά ως προς τη διορθωτική επιστολή για το 2015. Θα βρεθούν αυτά τα θέματα στο επίκεντρο των συζητήσεων και στη συνδιαλλαγή. Η Επιτροπή Γεωργίας θα εξετάσει τη διορθωτική της ε, τη διορθωτική αυτή επιστολή στην επόμενη τη συνεδρίαση, την Πέμπτη το πρωί, αν δεν κάνω λάθος και σίγουρα και στην ε, σχετική συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας ε, θα λάβει μέρος μια αντιπροσωπή και της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού. Φαντάζομαι η κυρία Σάμπαλ θα δώσει το παρόν και ίσως και άλλα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών στην μεθαυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ πάντως θερμά τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας που έλαβαν μέρος στη συνεδρίασή μας και ο κύριος Πίτερ Γιάρ που είναι ο εισηγητής για το θέμα αυτό δυστυχώς ε, δεν μπόρεσε να έρθει και ζήτησε συγγνώμη για την απουσία του. Περνάμε τώρα στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2014. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ζεράρντε Πρέ. για να μας παρουσιάσει τα διαδοχικά σχέδια διορθωτικών προπολογισμού που μέχρι στιγμής δεν ψηφίστηκαν, αλλά είπαμε σήμερα ότι θα κάνουμε μια ενδεικτική ψηφοφορία για αυτά. Κύριε Ντεπρέ, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είχαμε συμφωνήσει, υπενθυμίζω πρώτα την στρατηγική που έχουμε καθορίσει με λίγα λόγια με ομοφωνία οι πολιτικές ομάδες απεφάσισαν να ζητήσουν συμφωνία με το Συμβούλιο για το Σχέδιο Διορθωτικού Προϋπολογισμού 2014 πριν από την Συμφωνία για τον Προϋπολογισμό 2015. Δεύτερο, Κατά συνέπεια, αποφασίσαμε να συζητήσουμε τους ιδιορθωτικούς προϋπολογισμούς από τον 1, από τον 2 μάλλον, γιατί ο 1 έχει ήδη εγκριθεί, μέχρι τον 7. Αυτά στην προηγούμενη Ολομέλεια εγκρίθηκαν και σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 2 ώστε τα χρήματα που περιλαμβάνει αυτό το, αυτό το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού να μπορέσουν να εισέλθουν στον προπολογισμό. Τώρα, επειδή δεν θα έχουμε την ευκαιρία γιατί το Συμβουλίο δεν έχει τοποθετηθεί παρά μόνο για τον διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 2. Δεν έχουμε λοιπόν την δυνατότητα να ψηφίσουμε σε ολομέλεια θέση για τους υπόλοιπους draft amending budgets, αλλά θα επανέλθουμε στις 6 του μηνός, γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε και να τελειώσουμε στις 14 του μηνός. Θα μας τα πείτε βέβαια αυτά για το χρονοδιάγραμμα. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε την ευκαιρία να καταλήξουμε σε θέση της Ολομέλειας, επιθυμώ σήμερα να κάνουμε μια ενδεικτική ψηφοφορία για το σύνολο των εκθέσεων που υποβάλλω για τους διάφορους αυτούς διορθωτικούς προπολογισμού και που στο σύνολό του το νόημα λέει ότι αν τους πάρουμε όλους μαζί θέλουμε να ψηφιστούν όλοι μαζί, να εγκριθούν όλοι μαζί. Όσοι έχουν από το Συμβούλιο επίσης. Είχα την ευκαιρία ήδη να σας παρουσιάσω τον, ε, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαρθμών 3. Είναι αυτό το οποίο κατ' ουσία αυξάνει κατά 4 δισεκατομμύρια 700 εκατομμύρια το σύνολο των πιστώσεων πληρωμών και να χρησιμοποιήσουμε και το λεγόμενο contingency margin. Αυτό λοιπόν το draft amending budget που σας υποβάλλω και που περιλαμβάνεται και στην ημερήσια διάταξη έκθεση υπαριθμών 6, κινητοποίηση του περιθωρίου για πρόβλεπτα για το 2014, γιατί για να κινητοποιηθεί το περιθώριο αυτό χρειάζεται ειδική νομική πράξη. Προτείνω λοιπόν να εγκριθεί αυτή η νομική πράξη στο σημείο 6. Τώρα για τους 4 και 5 διορθωτικούς προϋπολογισμούς. Αυτοί σας έχουν ήδη υποβληθεί. Πάλι εκεί πρόκειται για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Δεν είναι δική μου εκθέση, είναι οι άλλες εκθέσεις. Και μένουν οι παριθμών 6 και 7 Σύντομα θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίω για τον υπαριθμόν 6, να παρουσιάσει το περιεχόμενο αυτών των δυο διορθωτικών προϋπολογισμών, ώστε όλοι να μπορέσουν να κατανοήσουν το εύρος τους και την σημασία τους. Αλλά πάντως αυτό που ζητώ είναι συνολική έγκριση αυτών των διορθωτικών προϋπολογισμών από τον αριθμό 2 έως τον αριθμό 7. Εσείς τώρα κυρία Καλβίνιο για τον αριθμό 6 πρώτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω και εγώ να μιλήσω αργά και με σαφήνεια, γιατί ο διορθωτικός προεπλογισμός υπαριθμών 6 είναι πάρα πολύ περίπλοκος και πάρα πολύ τεχνικός. Λοιπόν, ε, το σχέδιο διορθωτικού προεπλογισμού του υπαριθμών 6 κατ' ουσίαν αφορά την προσαρμογή των ιδίων πόρων κάτι το οποίο γίνεται έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικαιροποιήσουμε τα έσοδα του προεπλογισμού με βάση της, ε, την πραγματική εξέλιξη των ιδίων πόρων. Ε, φέτος λοιπόν είχαμε κάτι το θετικό. Είχαμε μεγαλύτερα έσοδα από τους δασμούς. Το αρνητικό ήταν ότι ήταν μικρότερα τα έσοδα από το ΦΠΑ. Και κατόπιν υπάρχει και ένα τρίο, τρίτο στοιχείο που έχει να κάνει με την προσαρμογή ε, του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος των διαφόρων κρατών μελών. Αυτή λοιπόν είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο και προκύπτει από μία σειρά συνεδριάσεων των στατιστικών υπηρεσιών των διαφόρων κρατών μελών. Είναι μία ανεξάρτητη διαδικασία που λαμβάνει η χώρα ανάμεσα στις στατιστικές υπηρεσίες και τη Eurostat. Εκεί εξετάζονται τα στοιχεία και τελικά καταλήγουν στο ότι υπάρχουν ε, τα τελικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την διαπίστωση των ιδίων πόρων. Πρέπει να σας πω ότι όλη αυτή η διαδικασία ε, και τα αποτελέσματα προκάλεσαν ε, αντιδράσεις ε, στα κράτη-μέλη, διότι η προσαρμογή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, κυρίως για τους ισολογισμούς του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Τώρα, ο λόγος ήταν ότι τα κράτη-μέλη έκαναν πολλές αναθεωρήσεις στα στοιχεία ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των ετών 2002 μέχρι το 2014. Και αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους, διότι βελτιώθηκε και η μέθοδος των διομπορών κατόπιν ε, σαν επιφυλάξεις που είχαν προκύψει από πλευράς Eurostat και πολλά άλλα. Εκείνο λοιπόν το οποίο προτείνουμε εμείς με τον διορθωτικό προϋπολογισμό, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 6 είναι καταρχήν να υπάρξει αύξηση των παραδοσιακών ιδίων πόρων κατά 420 εκατομμύρια έτσι ώστε να ε, φαίνονται καλύτερα τα αυξημένα έσοδα που έχουμε από τους, από τους δασμούς. Κατόπιν, 285 εκατομμύρια από το ΦΠΑ. Και τρίτον, ένα 9,8 δισεκατομμύρια για να υπάρξει αντιστάθμιση των επιπρόσθετων εσόδων που θα καταγραφούν στον προπλογισμό μέσα από την αυτόματη προσαρμογή του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Άρα δηλαδή για να είμαστε σαφείς, αν δεν τροποποιήσουμε τον υπαριθμό 6 μέχρι την 1η Δεκεμβρίου, τότε τα κράτη-μέλη θα αναγκασμένα στον ευρωπαϊκό προπλογισμό να καταβάλουν περίπου 9 δις ευρώ, κάτι το οποίο όμω δεν το χρειαζόμαστε τώρα, γιατί σας είπα έχουμε αρκετά έσοδα από τους ίδιους πόρους και από αυτά τα επιπρόσθετα έσοδα που λάβαμε φέτος αυτά θα προκύψουν από τον διορθωτικό προπλογισμό υπαρτιμών 4 και από άλλους. Κατόπιν τούτου αυτό το οποίο προτείνουμε είναι τα χρήματα αυτά να επανέλθουν στα κράτη-μέλη. Άρα δηλαδή αυτό είναι καλό, θετικό για τα κράτη-μέλη. Βεβαίως η σχετική εισφορά των κρατών μελών έχει τροποποιηθεί λόγω και της προσαρμογής στο καθάριστο εθνικού εισοδήματος. Ορισμένα κρατημέλη εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ευκαιρία και αναθεώρησαν προς τα επάνω το καθάριστο εθνικό εισόδημα, άρα δηλαδή έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στις ε, συνεισφορές ιδίων πόρων με βάση το καθάριστο εθνικό εισόδημα. Άρα δηλαδή το ποιο θα λάβει πίσω χρήματα και ποιο θα καταβάλει μεγαλύτερα ποσά στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και προφανώς συζητείται στο Συμβούλιο. Αλλά ο διορθωτικός προπολογισμός υπαριθμών 6 κατ' ουσίαν επιστρέφει κονδύλια στα κράτη-μέλη διότι δεν χρειαζόμαστε μεγαλύτερα έσοδα ως έχουν τα πράγματα τώρα. Τώρα, ο διορθωτικός προπολογισμό υπαριθμών 7 είναι πολύ διαφορετικός με την έννοια ότι έχει να κάνει με την κινητοποίηση του ε, Ταμείου Λεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σχέση με τις πλημμύρες στη Σερβία και την Κροατία το το Μάιο του 2013 και τις πλημμύρες ε, ε, που έλαβαν χώρα εφέτος ε, και έπληξαν σε μεγάλο βαθμό τη Σερβία και λιγότερο την Κροατία προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στην υποδομή, επίσης κατέστρεψαν πάρα πολλά νοικοκυριά. Και αφού συνέβησαν αυτά, μετά από δύο μήνες, το ίδιο επαναλήθηκε και στη Βουλγαρία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε εντελεχή εξέταση των αιτήσεων και από τα τρία κράτη-μέλη με βάση τους κανονισμούς που ισχύουν για το Ταμείο Λεγγύης και εμείς προτείναμε να κινητοποιηθεί το Ταμείο Λεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης να δοθεί στις χώρες αυτές το ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Σας ευχαριστώ. Votre, votre Η κυρία Μούντι ζήτησε το λόγο, γιατί φαίνεται υπάρχουν απορίες από την παρουσίαση που μας κάνατε. Σας ευχαριστώ. Όπως είπατε, η σχέση μας με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 6 είναι γνωστή και υπάρχουν όμως αντιδράσεις από το Συμβούλιο. Και συμφωνώ ότι το θέμα δεν είναι μόνο τεχνικό, επέκτησε και πολιτικές διαστάσεις, όλο και αυξανόμενες. Και η αποτυχία πολιτικής διαχείρισης ε, του θέματος επιδίνωσε την κατάσταση και παρεμπόδισε την έγκριση του σχεδίου διορθωτικού προπολογισμού υπ. 6 πολύ πιο γρήγορα. Πάντως ε, χαιρετίζω τις προτάσεις σας ε, για την ε, διόρθωση κατάστασης φέτος και την αποτροπή επανάληψη τέτοιου φαινομένου στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Δεπρέ. Κύριε Πρόεδρε, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα σε σχέση με τις ε, αντιπαραθέσεις ε, που δημιουργήθηκαν για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6, θα ήθελα να διαλευκάνω ορισμένα θέματα για να μην υπάρχουν αφησιμίες και παρεξηγήσεις. Καταρχήν, ως προς τη διαδικασία που μας οδήγησε στο ποσό που αναφέρεται στο έγγραφο. Καταρχήν δεν πρόκειται για πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για εργασίες της ε, ε, Eurostat σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Ε, από αυτές τις εργασίες προέκυψε ο υπολογισμός των ποσών για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα κάθε χώρας δεν είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η συνεννοήσεις της Eurostat με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες που κατέληξαν στη συγκεκριμένα ποσά για τα καθάριστα εθνικό εισόδημα. Ακούσαμε τις αντιδράσεις ενός κράτους μέλους που το κακόμερο θα πρέπει να πληρώσει ενώ άλλοι θα λάβουν επιταγές. Καταρχήν υπάρχει δυνατότητα για ένα κράτος να αποφύγει τη πληρωμή συμπληρωματικού ποσού. Γιατί υπάρχει αυτό το, αυτή η κατάσταση σήμερα. Και ποιες είναι οι νομικές και δημοσιονομικές συνέπειες είτε καθυστέρησης της καταβολής αυτής της συμπληρωματικής πληρωμής είτε της αποφυγής. Και τρίτη ερώτηση. Και παρακαλώ δώστε μου μια ξεκάθαρη απάντηση. Είναι σαφές ότι με την έγκριση των σχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών 2-7 τα κράτη-μέλη θα επωφεληθούν ε, όλα. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη που, θα, που καλούνται να καταβάλουν θα πληρώσουν λιγότερο, ενώ αυτά που θα λάβουν ποσά θα επωφεληθούν περισσότερο. Θα ήθελα να το διευκρινίσουμε. Κύριος Σνότ, ευχαριστώ. Καταρχήν είναι σαφές ότι το ζήτημα αυτό έχει μείζωνα πολιτική σημασία και είναι ιδιαίτερα επίκαιρο αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί ο αντίκτυπο για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ σημαντικότερο από ό,τι οι επιπτώσει σε άλλα κράτη-μέλη ακόμη και με το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 6, μιλάμε για πάνω από 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ που καλείται το, Ευρωπαϊκό, το Ηνωμένο Βασίλειο συγγνώμη, να καταβάλει. Και δημιουργήθηκε πραγματικό σοκ με την είδηση αυτή όταν ξέσπασε. Ε, και φαίνεται ότι ο Ντέβιτ Κάμερον δεν είχε ιδέα για το τι τον περίμενε. Ερωτώ λοιπόν, θα έπρεπε να γνωρίζει η Βρετανική κυβέρνηση ότι κάποια στιγμή θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον ποσά. Ή γιατί κατα... καταλήφθηκαν όλοι εξαπίνης. Όφυλα να γνωρίζουν κάτι τέτοιο. Εκτός μικροφώνου το σχόλιο, θα ήθελα και μια επίσημη απάντηση. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για αυτή την τεράστια διαφορά. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο πληρώνει τόσο περισσότερα από ό,τι άλλα κρατημέλη. Βέβαια είπατε ότι οφείλεται στην αναθεώρηση των στοιχείων για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα που έκανε η Eurostat. Γιατί όμως οι διορθώσεις για τα άλλα κρατημέλη είναι σχετικά μικρές, ενώ για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι τόσο υψηλές. Ε, το η Ολλανδία έχει 642 εκατομμύρια που είναι από τα ψηλότερα ποσά, αλλά τα 2,1 δισεκατομμύρια του Ηνωμένου Βασιλείου ξεπερνούν κατά πολύ όλε τι ε, υπόλοιπε χώρε. Άλλωστε ο Ντέβιτ Κάμερον δήλωσε ότι δεν πρόκειται να πληρώσει την 1η Δεκεμβρίου. Ε, Προφανώ θα υπάρξουν συνέπειε από μια τέτοια άρνηση. Έχουμε και το άρθρο 11 του κανονισμού 1150 του 2000 η άνηση πληρωμής ενεργοποιεί τόκους υπερημερίας και μάλιστα κάθε μήνα που περνά οι τόκοι αυτοί αυξάνονται. Ακούγουμε στο, και διαβάζουμε στο Βρετανικό τύπο ότι θα γίνουν διαπραγματεύσεις για την διόρθωση του ποσού. από τη μια ακούμε ε, ότι θα γίνουν διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του ποσού, απ' την άλλη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταβάλει και επιπλέον πρόστιμα αν αρνηθεί να πληρώσει. Ποια είναι η αλήθεια λοιπόν για την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Καλβίνιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις ε, ερωτήσεις. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν και γιατί ισχύουν. Ο κανονισμός υπαριθμών 50, ε, στον οποίο αναφερθήκατε, αποτελεί το βασικό κανονισμό ε, σε σχέση με την ίσπραξη ιδίων πόρων. Και ο κανονισμός υπαριθμών 50 11.50 είναι πολύ λεπτομερής και περιγραφικός και ε, αναφέρεται συνέχεια στο τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μην υπάρχει, κανένα περιθώριο διακριτικής ευκαιρίας ε, σε επίπεδο επιτροπής ή κρατών μελών να αποφασίσουν κατά πόσον θα καταβάλουν τα ποσά ή όχι. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει λόγος που γίνεται ή τουλάχιστον δύο λόγοι. Δηλαδή, καταρχήν, γιατί πρέπει ο ε, προϋπολογισμός να είναι πάντα ισοσκελισμένος, να υπάρχει η σαφήνεια κατα ποσον τα καταβαλουν τα ποσα η οχι και αυτο γινεται γιατι υπαρχει λογος που γινεται η τουλαχιστον δυο λογοι δηλαδη καταρχην γιατι πρεπει ο προυπολογισμος να ειναι παντα ισοσκελισμενος να υπαρχει η οτι τα κράτη-μέλη θα πληρώσουν και μάλιστα μερικά εξ αυτών πράγματι το πράττουν. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει και εκείνα να είναι σίγουρα ότι θα αντιμετωπίζονται με ίσους όρους, ότι δεν θα υπάρχει ειδική μεταχείριση κάποιων κρατών μελών. Και γι' αυτό το λόγο οι κανόνες είναι σαφείς και λεπτομερείς. Η όλη διαδικασία αναφέρεται ε, στη συγκέντρωση των δεδομένων που κατά κανόνα μέσα Οκτωβρίου αποκτάμε τα τελικά στοιχεία που, έχουν, ε, που για, την, ε, για τον υπολογισμό των συνεισφορών. Ο υπολογισμός γίνεται κάθε χρόνο, υπάρχουν κάθε χρόνο αλλαγές, φέτος όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί τα κράτη-μέλη εκμεταλλεύτηκαν αυτή την αλλαγή που υπάρχει με τους νέους στατιστικούς κανόνες. Ε, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό και αναθεώρησαν το ακαθάριστο εθνικό τους εισόδημα. Και ορισμένοι εξ αυτών το αναθεώρησαν σημαντικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αλλαγές ήταν μεθοδολογικής φύσεως, σε άλλες περιπτώσεις ε, εντάχθηκαν ε, όλα αυτά στις δραστηριότητες Πάντως, ε, στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, η σημαντικότερη αλλαγή είναι το ότι ε, συμπεριλαμβάνονται οι δωρές ε, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Η διαδικασία λοιπόν είναι ίδια, ακολουθείται κάθε χρόνο και βασίζεται στη δουλειά των ε, Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών. Συμφωνώ όμως ότι αυτά τα στοιχεία, το καθάριστο εθνικού εισοδήματο είναι σωστά για το θέμα των ιδίων πόρων και πρέπει να είναι σωστά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναμίχθηκε σε αυτή τη διαδικασία για λόγους ε, στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Εμείς ε, είχαμε να τηρήσουμε αυστηρές προθεσμίες γιατί κανονικά αυτοί οι υπολογισμοί γίνονται όσο πιο πολύ στο τέλος του έτους έτσι ώστε να μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Η αναθεώρηση λοιπόν έγινε στα μέσα Οκτωβρίου. Στις 17 Οκτωβρίου υποβάλαμε τα αναθεωρημένα στοιχεία σε όλα τα κράτη-μέλη. Το ερώτημα κατά πόσο μπορεί κάποιο κράτος μέλος να μην πληρώσει, η απάντηση είναι όχι. Ο κανονισμός λέει ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να πληρώσουν μέχρι την 1η Δεκεμβρίου. Δεν υπάρχει ε, καμία διακριτική ευχαίρεια ως προς την προθεσμία, ούτε ως προς το ποσό και τελικά αν η πληρωμή δεν γίνεται μέχρι την 1η Δεκεμβρίου δεν υπάρχει και διακριτική ευχαίρεια ε, να μην καταβληθούν οι τόκοι των ε, προστήμων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του 1150. Τώρα, κατά πόσον πλήττεται ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, με απόλυτους όρους ναι, σχετικά όμως όχι. Άλλα κράτη-μέλη έχουν μεγαλύτερες διορθώσεις ως ποσοστό το καθαριστο εθνικου εθνικού εισοδήματο, γιατί υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη που καταβάλουν περισσότερα από τα Ολλανδία, Μάλτα, Κύπρος, Ελλάδα. Αυτά είναι τα μικρά και εκεί η διόρθωση που γίνεται είναι πολύ μεγαλύτερη για τον προϋπολογισμό τους. Και θα ήθελα ολοκληρώνοντας να πω το εξής, ότι η Κομισιόν δεν έχει κανένα περιθώριο να αναδιαπραγματευτεί τα ποσά. Υπάρχει ο κανονισμός και η απόφαση του δικαστηρίου και σας λέω ότι η Κομισιόν δεν είναι ότι μπορεί να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις τα κράτη-μέλη για να αποφασιστεί το κατά πόσον ένα κράτος θα πληρώσει ή όχι. Αυτά λοιπόν προβλέπονται στον κανονισμό. Και τώρα πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτά να ξανασυμβούν. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, διότι όταν συντάχθηκε ο κανονισμός τότε δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε απρόβλεπτες καταστάσεις που μπορεί να προκύψει μια φορά στα 15 χρόνια. Άρα δηλαδή Πρέπει να δούμε πώς θα τα αποφύγουμε όλα αυτά στο μέλλον. Πάντως, κατά τις επόμενες εβδομάδες, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο κανισμός δεν αφήνει περιθώριο ελιγμών για να ε, ανταποκριθεί κανείς σε, σε πολιτικές καταστάσεις που έχουν προκύψει με τεχνικά μέσα. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να διατυπώσω την άποψή μου. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, ερωτήσεις, ε, να ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή εξ αρχής ε, ζητώ συγγνώμη αν οι ερωτήσεις μου κρυθούν αφελείς. Εγώ είμαι νέος σε αυτή την Επιτροπή και δεν έχω καταλάβει καλά πώς ακριβώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός ο οποίος οδήγησε στον, στο σχέδιο διορθωτικού προβλησμού στο υπαριθμόν 6. Ε, αν κάνω λάθος, συνάλλως να με διορθώσει. Έχω δίκιο στο τα κράτη-μέλη

αναθεώρησαν ε, το ακαθάριστο εθνικό εισόδημά τους με βάση τους ε, νέους κανονισμούς. Εάν αυτό ισχύει, τότε κατά τη δική μου άποψη αυτό είναι ανόητο. Διότι αυτή τη στιγμή ζητάμε είτε περισσότερα χρήματα είτε λιγότερα χρήματα από τα κράτη-μέλη με βάση ενός νέου υπολογισμού του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος που όπως στην περίπτωση της Ιταλίας εκεί κατά τον υπολογισμό συμπεριλαμβάνεται και η παραοικονομία και όπως είπα είπατε κι εσείς προηγουμένως, ε, ε, συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα από τα ναρκωτικά, από την πορνεία, αυτά δηλαδή που μπαίνουν στην παραοικονομία. Αυτά όμως αντιβαίνουν στην ίδια την αρχή του υπολογισμού του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, γιατί αυτό το χρησιμοποιεί κανείς για να υπολογίσει τον πλούτο μιας χώρας. Και βλέπουμε ότι εδώ εμπίπτουν όλες οι δραστηριότητες οι οποίες αποδίδουν φορολογικά εισοδήματα. Η παραοικονομία εξορισμού αυτή δεν αποδίδει φορολογικά έσοδα. Άρα δηλαδή σας λέω ότι εδώ πρόκειται για μία αντίφαση και ίσως μπορείτε λιγάκι να μου εξηγήσετε περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Εμείς ζητάμε επιπρόσθετα κονδύλια με βάση τεχνητούς υπολογισμούς οι οποίοι κατά την άποψή μου είναι παντελώς παραπλανητικοί ή αν θέλετε ο νέος υπολογισμός οφείλεται στο ότι οι εισφορές με βάση το καθάριστο εθνικό εισόδημα υπολογίζονται στις αρχές του έτους και κατόπιν στο τέλος του έτους να έχουν αλλάξει κάπως τα στοιχεία προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Δεν ξέρω, η Ιταλία ας πούμε στις αρχές του έτους ε, μπορεί να έχει ένα χ υπολογισμό και στο τέλος του έτους να προκύπτει ότι ε, το 100 που είχε υπολογιστεί στην αρχή έχει γίνει 104. Θα ήθελα λιγάκι να μου τα διευκρινίσετε αυτά για να τα καταβάλω. Επίσης, από το 2000 μέχρι το 2013. Νομίζω ότι αυτό το χρονικό διάστημα αφορά και την περίοδο που μπήκαν οι νέοι υπολογισμοί. Γι' αυτό λοιπόν, ε, φαντάζομαι, γι' αυτό επελέγει αυτό το χρονικό διάστημα. Επίσης, μπορείτε να μου πείτε κατά πόσον μπορούν να υπολογίζονται μικρότερα χρονικά διαστήματα για να μην συμβαίνει αυτό που συνέβη παραδείγματος χάρη με το Ηνωμένο Βασίλειο, να προκύπτουν τόσο μεγάλα ποσά. Και η τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω αφορά αυτό που είπατε ότι τα κράτη-μέλη επέλεξαν ε, να εποφεληθούν από ε, το ε, υπαριθμών 10 για τον επανυπολογισμό. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν μια επιλογή των κρατών μελών, ίσως για να κάνουν κάποιες εξοικονομήσεις σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα. Πάντως ε, στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι αυτοπυροβολήθηκαν όσον αφορά τουλάχιστον στον υπολογισμό των συνεισφορών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις γιατί κατά την άποψή μου όσον αφορά το σχέδιο του διορθωτικού προϋπολογισμού των υπαρτμών 6 το θέμα δεν είναι σαφές. Ποιος θέλει, τι είναι η υπετιότητα, η υπετιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών που προσπάθησαν να επωφεληθούν από ένα λογιστικό τέχνισμα για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα, αλλά τελικά την πάτησαν, α το πούμε απλά, γιατί βρέθηκαν να είναι αναγκασμένοι να καταβάλουν μεγαλύτερα ποσά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Στονάνο. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Μερικοί μάλιστα από τις εφημερίδες μάθαμε το βρετανικό πρόγραμμα με τα περίφημα αυτά δύο δις ε, που καλείται να καταβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το έργο της Eurostat. Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν σαφείς κανόνες, όπως φαίνεται, που μάλιστα εφαρμόζονται από ανεξάρτητο οργανισμό, είναι δυνατό να υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να γίνουν σεβαστοί και να εφαρμοστούν οι κοινοί μας κανόνες. Τώρα βέβαια εδώ φαίνεται ότι αγγίζουμε τα όρια του συστήματος των ιδίων πόρων με τη μορφή που έχει σήμερα τουλάχιστον. Και το είπαμε επανειλημμένως και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι τώρα ξεκινάει αυτή η συζήτηση. Και το θέμα της παραοικονομίας με ενδιαφέρει ε, ιδιαίτερα. Σε ποιο επίπεδο παραοικονομίας σταματάμε. Γιατί η αλληλέγγυη και κοινωνική οικονομία δεν είναι παραοικονομία. Είναι ανοιχτή, δημόσια, εμφανής και συμπεριλαμβάνεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα. Η παραοικονομία όμως είναι πραγματικά παράνομη οικονομία. Οπότε πώς συνυπολογίζεται. Θα πρέπει να έχουμε κοινού κανόνες για τον προσδιορισμό της και τη ρύθμιση της. Ο κύριος Τάραντ. Σας ευχαριστώ. Ό συνήθως η ομάδα μας συμφωνεί με τις προτάσεις του εισηγητού. Έχω κάποιες επιφυλάξεις όμως για την τακτική μας σε ό,τι αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 6. Γιατί αν το εγκρίνουμε τώρα θα δείξουμε υπερβολική καλή θέληση προς το Συμβούλιο που μας ε, είχε τις ε, μήνους, μήνες ολόκληρους ε, με ανεδαφικά νομικά επιχειρήματα προκειμένου μόνο και μόνο για να, να κολλησιεργήσει και να καθυστερήσει την υιοθέτηση του σχεδίου. Και τώρα να αποκρισταλώσουμε εμείς τη θέση μας πολύ πριν από το Συμβούλιο, ουσιαστικά θα παίξουμε το παιχνίδι του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο θα, θα ευνοήσουμε και όχι τους, ε, τα άλλα μέρη της διαδικασίας. Πέραν τούτου συμφωνώ με την πρόταση. Ε, δεν συμφωνώ συγγνώμη την πρόταση για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Ε, uh, yes, Ο κύριος Όλμπριχτ. Είμαι ο σκιώδης ε, εισηγητής για όλα αυτά τα σχέδια διορθωτικού προϋπολογισμού και θα ήθελα να πω ότι εμείς φυσικά θα στηρίξουμε τον εισηγητή μας και είναι σημαντικά τα συμπεράσματα της συζήτησης, ότι θα πρέπει να εμείνουμε στις αρχές μας, ότι θα πρέπει να κρατήσουμε αδιέρετο το πακέτο με τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών. Και παρά τα προβλήματα και τις επιφυλάξεις που έχουμε για τη μεθοδολογία, που έχει συμφωνηθεί από τα κράτη-μέλη, από ό,τι ξέρω, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν επί της μεθοδολογίας. εφαρμόστηκε, και τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά για τα κράτη-μέλη, αλλά δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης πλέον η μεθοδολογία. Και δεν θα πρέπει το σχέδιο προπολογισμού υπαριθμών 6 να το κρίνουμε ω στοιχείο που μπορεί να καταστρέψει το πακέτο. Θα πρέπει να μείνουμε στην αρχή να κρατήσουμε το πακέτο ακέραιο Όπω πρότεινε ο εισηγητή, και να ξεκινήσουμε τη συνδιαλλαγή για τα σχέδια διορθωτικού προπολογισμού πρώτα το 2014 και μετά να περάσουμε στον προπολογισμό του 2015. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό είναι και το συμπέρασμα που έβγαλα εγώ από τη συζήτηση. Ότι οι συζητήσει μα για το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 6 δεν αλλάζουν επί τη ουσία στη θέση μα ω προ το πακέτο των διορθωτικών προπολογισμών. Ο κύριο Δεπρέ. Νομίζω ότι όλοι έχουν τοποθετηθεί έτσι, δεν είναι κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πράγματι, εκτός αν ίσως η κυρία Καλβίνιο θέλει να επανέλθει. Για να απαντήσει στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις που τέθηκαν. Και αμέσως μετά θα σας δώσω το λόγο για να ολοκληρώσετε κύριε ε, Ντεπρέ. Η κυρία Καλβίνιο. Ευχαριστώ και πάλι Πρώτα λησμόνησα να αναφέρω την Ιταλία που είναι η άλλη χώρα η οποία θίγεται από την θετική συμβολή, η Δεν χρησιμοποίησαμε τους νέους κανόνες 2010 για το, το ΣΕΚ, 2010. Οι, οι ίδιοι πόροι, οι αποφάσεις του τους ίδιους πόρους εγκρίνονται αναχώρα μέλος, στις χώρες μέλη δηλαδή. Χρησιμοποιούμε ακόμα λοιπόν το ΣΕΚ 95. Όμως, επειδή οι χώρες μέλη περάσαν ήδη στο ΣΕΚ 2010, ίσως έχουν λάβει την ευκαιρία για να συζητήσουν διάφορες αλλαγές στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημά τους. Στον τρόπο υπολογισμού δηλαδή. Δεν γνωρίζω ακριβώ τι έχουν κάνει τα εθνικά στατιστικά γραφεία, αλλά ο υπολογισμό έχει βασιστεί στα δεδομένα που έχουν υποβάλει οι Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες. Εμείς διαπραγματευθήκαμε και με την Ευρωστάτη για ορισμένες επιφυλάξεις, αλλά τις χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά για τον υπολογισμό των ιδίων πόρων. Τώρα, μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει συντομότερη περίοδο. Η συνήθις περίοδος είναι 9 ετών, εκτός αν υπάρχουν επιφυλάξεις. Οπότε οι υπολογισμοί μπορεί να καθυστερήσουν κι άλλο. Πάλι, η χρήση των δεδομένων αυτών απορρέει από την διαδικασία αυτή που κινείται μεταξύ των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών. Εδώ βάζω και ένα σχόλιο εντός παρενθέσεων. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ακαιρεότητα της ε, στατιστικής διαδικασίας, διότι είδαμε τα αποτελέσματα όταν προσπάθησαν να, κάνουν, να πολιτικοποιήσουν την δράση των στατιστικών υπηρεσιών. Εμείς ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα να παραμείνουν ανεξάρτητες οι στατιστικές υπηρεσίες. Τώρα για τους κοινού κανόνες. Οι κανόνες είναι κοινοί, τα αυτοί που δηλαδή ε, εφαρμόζουμε εμείς, αλλά επανεξετάζεται ο τρόπος ερμηνείας των κανόνων. Σημαντικό επίσης να μην λησμονεί κανείς ότι ο παρόν διορθωτικός προϋπολογισμός, ο υπαριθμών 6 δηλαδή, δεν σημαίνει παραπάνω χρήματα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δεν σημαίνει παραπάνω χρήματα για τις Βρυξέλλες, να το πω έτσι αποτελεί εκ νέου εξισορρόπηση μεταξύ των χωρών μελών. Και κάτι που είπαν ορισμένα από τα μέλη σας είναι ότι ορισμένε χώρε μέλη θα πληρώσουν περισσότερα και άλλε θα λάβουν περισσότερα. Πρόκειται λοιπόν για εξισορρόπηση μεταξύ των χωρών μελών. Το συνολικό πακέτο τώρα των διορθωτικών προπολογισμών που ζήτησε ο κ. Ντεπρέ έχει θετική έκβαση. Συνολικά δηλαδή πλεόνασμα 87,5 εκατομμυρίων ευρώ που θα καταβληθούν στις μέλη. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό απαντώ στις διάφορες ερωτήσεις που θέσατε. για αυτό το ζήτημα του DAB 6, το Διευθυντικού 6. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντεπρέ για να μπορέσει να ολοκληρώσει. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε αυτό το πακέτο των δημοσιονομικών διορθώσεων, αλλά τη στιγμή που θα ψηφίσουμε. Κύριε Ντεπρέ, εσείς. Το ΣΕΚ είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών, σημειώνει η Κοιτάξτε, δεν είναι σωστό να αλλάζει κανείς στρατηγική την τελευταία στιγμή που πάει να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο. Διότι το πρόβλημα είναι ότι αποδυναμώνει κανείς την θέση του ο ίδιος. Γιατί αλλάζει και η σύνθεση της ομάδας. Ας διατηρήσουν τις θέσεις τους οι συναδελφοί μου, ότι δηλαδή δεχόμαστε το σύνολο των διορθωτικών προϋπολισμών από τον αριθμό 2 έως τον αριθμό 7. Και όποιο και αν είναι το περιεχόμενο του σχεδίου διορθωτικού προϋπολισμού 6. Δεν υπήρξε σφάλμα ούτε από το Κοινοβούλιο ούτε από την Κομισιόν σχετικά με το ποσό. Οι χώρες μέλη καθόρισαν το ύψος του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωστάτ. Σε ποια βάση το έπραξαν δεν γνωρίζω. Ίσως ορισμένες χώρες μέλη ήθελαν να δείξουν με τον τρόπο τους ότι έχουν υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη από άλλες. Τόσο το καλύτερο για αυτές. Να πω λοιπόν στον συνάδελφό μου, τον πρασίνων εδώ πίσω μου, σας παρακαλώ να μην καθυστερήσουμε την ψηφοφορία ούτε να καταψηφίσετε αυτόν τον διορθωτικό 6. Διότι ποιο μήνυμα θα δώσουμε να το κάνουμε αυτό. Κάνα θετικό μήνυμα. Κάνας δεν έχει βάλει πρόβλημα. Βάζουμε εμείς πρόβλημα τώρα. Αν, δεχτούμε, αν δεν δεχτούμε το αποτελέσμα των υπολογισμών, αλλάζουμε στο τόπεδα. Αντί να είμαστε λοιπόν, να συμπαραταχθούμε με την πλειονότητα των χωρών μελών που θα λάβουν περισσότερα, δίνουμε λάθος μήνυμα αν διστάσουμε. Και θα ήταν επί της ουσίας βαρύ σφάλμα. Αλλά και στο επίπεδο της τακτικής πάλι θα ήταν λάθος απέναντι στο Συμβούλιο. Με κάθε λοιπόν δυνατή πειθό σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε στην βάση των προσανατολισμών που έχουμε ήδη δεχτεί. Μάλιστα, θα δούμε σε λίγα λεπτά, κύριε Ντεπρέ, όταν θα αρχίσουν οι ψηφοφορίες και ιδίω η πρώτη ενδεικτική ψηφοφορία για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον περίφημο 6, δεν έχει συνέπεια στο δημοσιονομικό υπόλοιπο που μας απασχολεί. Πρόκειται για πρόβλημα μεταξύ των χωρών μελών και εάν εν τέλει υπάρξουν κάποιες διαπραγματεύσεις οι χώρες οι οποίες θα είναι δικαιούχοι θα περιμένουν διότι οι άλλες δεν θα καταβάλουν αμέσως τα σχετικά ποσά. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ποιο είναι το νόημα του μηνύματός σας. Το πακέτο δεν πρέπει να αφήσει κανέναν διορθωτικό προϋπολισμό απ' έξω. Αν λοιπόν συμφωνείτε να προχωρήσουμε τώρα στους δημοσιονομικούς κανόνες για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, θέμα όπου η είναι η κυρία Γκρέσλε και να δώσουμε και τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας φωτίσει για το σχέδιο αυτό. Ο κύριος Ερικ Παραντή παρακαλώ να λάβει τον λόγο. Oui, merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια και μου δίνετε την ευκαιρία, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η καταπολέμηση, η πάταξη της απάτης ε, είναι πρωταρχικός στόχος και της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και στις επιστολές ε, ανάθεση καθηκόντων που έστειλε ο πρόεδρος Γιούνκερ σε όλους τους επιτρόπους περιλαμβάνεται το θέμα της πάταξης της απάτης ε, ως ύψητη προτεραιότητα και μάλιστα τα χαρτοφυλάκια των προϋπολογισμών της απαλλαγής ε, και της Όλαφ συγκεντρώνονται ε, στις αρμοδιότητες της Αντιπρόεδρου Τζόρτζεβα. Έτσι θα επιτύχουμε συνέργειες ε, στο δημοσιονομικό τομέα. Μία έγκαιρη ανείχνευση και αποκλεισμό των αναξιόπιστων ε, εμπορικών παραγόντων ήταν ε, ο λόγος για τον οποίο υποβάλαμε την πρόταση. Και φυσικά ε, διευρύνονται οι διερευνητικές δυνατότητες της Όλαφ. Βέβαια το σύστημα που προτείνουμε γνωρίζουμε ότι θα έχει επιπτώσεις στους οικονομικούς τελεστές και ίσως και στην οικονομική τους κατάσταση αλλά και την υπόλοιψή τους στην εμπορική. Θα πρέπει λοιπόν για να αποφύγουμε δυσμενή συνέπειε να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ τη προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση αφενό και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των οικονομικών τελεστών αφετέρου. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο συμπεριλάβαμε στην πρότασή μα διαδικαστικά εχέγγυα ώστε ο οικονομικό τελεστή να έχει τη δυνατότητα ακρόασης. Θεσπίσαμε την αρχή της αναλογικότητας και προτείναμε και την σύσταση ενός πάνελ, κεντρικού πάνελ, που θα εξετάζει όλες τις υποθέσεις. Έχουμε ένα κεντρικό φορέ λοιπόν. Έτσι θεωρώ ότι βρήκαμε την ισορροπία μεταξύ της ε, επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και της ε, διατήρησής τους και της δημοσιότητάς τους και το θέμα της δημοσιότητας των στοιχείων των αποκλεισμένων οικονομικών τελεστών. Και μάλιστα ο δεδομένων ε, μας ζήτησε να μην δημοσιεύουμε τις πληροφορίες αυτές για, τα, για τους ιδιώτες αλλά εμείς προτιμούμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της ε, διεθνούς διαφάνειας και να δημοσιεύουμε το σύνολο των πληροφοριών, είτε αφορούν πρόσωπα, είτε οργανώσεις. Και μάλιστα τον Νοέμβριο περιμένουμε και την επίσημη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Φροντίζουμε στην πρόταση να μην επηρεάζει που δεν είναι την υποχρέωση της Όλαφ για σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις ε, διαδικασίες έρευνας που ξεκινά. Και φυσικά προστατεύουμε και τους πληροφοριοδότες, τους καταγγέλλοντες, τους whistleblowers όπως λέμε στα αγγλικά. Με την πρότασή μας ε, συμπεριλαμβάνουμε στο δημοσιονομικό κανονισμό και θεσμοθετούμε τη συνεργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Όλαφ για την θέσπιση συντηρητικών και ασφαλιστικών μέτρων για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Και φυσικά λαμβάνεται υπόψη και ο κανονισμό της Όλαφ σε ό,τι αφορά την υποχρέωσή της να ενημερώνει αμελητή το θεσμικό όργανο για το οποίο έχουν ξεκινήσει ε, έρευνες την ενημέρωση της ανάγκης λήψης ασφαλιστικών συντηρητικών μέτρων. Και επίσης ενημερώνει ε, και το θεσμικό όργανο σε περίπτωση που αποφασίσει τη λήψη τέτοιων μέτρων. Θα ήθελα να να προσθέσω ότι η πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτυχε θερμής υποδοχής, ιδιαίτερα από τη διεθνή διαφάνεια, που μας έθεσε κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις κυρίως για τη σύνθεση του κεντρικού πάνελ που θα αποφασίζει τον αποκλεισμό ενός οικονομικού τελεστή. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που περιλαμβάνονται στο διατακτικό τμήμα, στο, στο δημοσιονομικό κανονισμό και στους εφαρμοστικούς κανόνες και ένα τμήμα που θα είναι εσωτερικό και θα αφορά απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά την κριτική για τον αποκλεισμό ε, και την αναφορά στην αιτιολογία της σύγκρουσης συμφερόντων. Δεν αποκλείεται η σύγκρουση συμφερόντων από τον κατάλογο των λόγων που οδηγούν σε αποκλεισμό. Και ο δημοσιονομικός κανονισμός, αλλά και το εσωτερικός κανονισμός ε, περιλαμβάνουν διατάξεις για να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων των ευρωυπαλλήλων. Σε περίπτωση κατεξαίρεση που θα έχουμε έναν ευρωυπάλληλο που θα είναι ταυτόχρονα και μέλος ενός διοικητικού συμβουλίου ή οργάνου διαχείρισης του οικονομικού τελεστή που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και που διαπράττει απάτη ή κάποια παρατυπία και ο δημοσιονομικός κανονισμός και το καθεστώς, ε, ο κανονισμός εταιρικής λειτουργίας προβλέπει μέτρα για αποκλεισμό αυτού του ευρωϊπαλλήλου ε, από την κρίση του οικονομικού τελεστή που μπορεί να έχει κάποια διαπλεκόμενα με τον ευρωϊπάλληλο. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό του σοβαρού επαγγελματικού σφάλματος. Η προσπάθεια επηρεασμού της διαδικασίας ε, λήψης αποφάσεων από την ε, αρχή ανάθεσης ε, ή απόπειρα απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών κατά τον διαγωνισμό. Νομίζω ότι και στα θέματα αυτά η έννοια της σύγκρουση φερόντων λαμβάνεται υπόψη. Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε ιδιαίτερα συζητήσει με τα κράτη-μέλη και μάλιστα εξετάσατε το σχετικό κείμενο ήδη μία φορά και περιμένουμε το σχέδιο έκθεση κυρία Γκρέσλε για να περάσει το θέμα στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων και μετά την οριστικοποίηση της έκθεσης να περάσουμε στους τριμερείς, στη διαδικασία των τριμερών διαλόγων. Τώρα, για τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη κυρίως ανησυχούν για τη γραφειοκρατία, για το επιπλέον γραφειοκρατικό άχθος που θα προκαλέσει υποχρέωσή τους ε, να αναφέρουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες παρατυπίες που επηρεάζουν οι ατασταλείς που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Πιστεύω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταφέρει να πει στα κρατη να δεχτούν αυτή την υποχρέωση κοινοποίηση, γιατί έτσι θα αυξήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, κυρίως της Όλαφ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών και θα σημειώσουμε πρόοδο στην καταπολέμηση της απάτης. Η πρόταση, η πρότασή μας, επαναλαμβάνω, έτυχε σχετικά θετική υποδοχή στην Επιτροπή Προπολογισμού από τα κράτη-μέλη και ελπίζω και η δική σα Επιτροπή Προπολογισμού να, τεχει, να επιφυλάξει την ίδια θετική υποδοχή. Κύριε Γκρέσλερ, τι λέτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μερικές φορές διαρωτόμαστε πού βρισκόμαστε ακριβώς. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την παρουσίαση. Πρόκειται για μια τράπεζα δεδομένων και θέλω να το εξηγήσω αυτό στους συναδέλφους. Ε, πρόκειται για μια τράπεζα δεδομένων κυρίως για όλους εκείνους οι οποίοι στο πλαίσιο διαδικασιών ε, προκήρυξη αγωνισμών εξαπάτησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα είδος μαύρου καταλόγου και η ιδέα που διέπει αυτή την τράπεζα δεδομένων είναι ότι να μην είμαστε αναγκασμένοι κάθε φορά να επιβραβεύουμε τους απαταιώνες. Αυτή η ιδέα είναι πάρα πολύ καλή. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί δεν λειτουργεί αυτή η ιδέα στην πράξη. Εγώ λοιπόν εδώ και 8 χρόνια ασχολούμαι περίπου με αυτή την τράπεζα δεδομένων και Ήδη κατά την πρώτη αναθεώρηση το 2006 Κατά το 2006 ασχολήθηκα με αυτή την τράπεζα δεδομένων και πραγματικά ήρθα σε έντονη αντιπαράθεση με τα κράτη-μέλη. Τότε είχαμε τον τριμερή διάλογο που λεγόταν βέβαια κάπως αλλιώς και αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο. Καταρτήσαμε αυτή την τράπεζα δεδομένων και σε αυτήν όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μόνο μία περίπτωση. Όχι γιατί δεν είχαμε περιπτώσεις, απλά γιατί δεν λειτουργήσε η τράπεζα δεδομένων. Τώρα λοιπόν αντιμετωπίζουμε την εξή πρόκληση. Πώς μπορούμε να έχουμε μία τράπεζα δεδομένων που να λειτουργεί. Νομίζω ότι αυτό είναι προς όφελος όλων μας. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τα ενωσιακά κονδύλια από απάτες και πώς είναι δυνατόν να μην επιβραβεύουμε εκείνους οι οποίοι έχουν ήδη λάβει κάποια κονδύλια και εξαπάτησαν. Εγώ ασχολούμαι με επιδοτήσει όπου μια οργάνωση που εξαπάτησε την Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε εκ νέου και πάλι κονδύλια. Αυτή λοιπόν η τράπεζα δεδομένων είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση και ξέρετε κύριε Παραντή, εγώ τελικά δεν έχω καταλήξει στο κατά πόσον αυτό που προτείνετε εσεί θα λειτουργήσει ή όχι. Οι συνάδελφοι που είναι νέοι συνάδελφοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνε που και εμεί. Ήδη δεν τους εφαρμόζουμε. Το ότι βέβαια δεν τους εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη, αυτό το ξέρουν όλοι, αλλά υπάρχουν και κανόνες που δεν τις εφαρμόζουν οι ίδιες οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράδειγμα, ακριβώς αυτή η Τράπεζα Ενδομένων, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφαρμόζει τους κανόνες που έχει ήδη αθεσπίσει, διότι το πρόβλημα ήταν τόσο μεγάλο που θα έπρεπε πριν συσταθεί αυτή η τράπεζα δεδομένων να υπάρχουν ήδη κάποιες αποφάσεις. Ακόμα και όταν υπάρχουν όμως δεν ενημερώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δαπανίσαμε πάρα πολύ χρόνο για αυτή την τράπεζα δεδομένων και τελικά αποδείχθηκε μία νοησία κατά το Τώρα πρέπει να βρούμε κάτι καλύτερο. Πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι σίγουρη ε, κατά πόσον αυτό που υπάρχει είναι ευρύθμο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι ρύθμιση υπάρχει πλέον ευκαιρία να βελτιώσουμε ορισμένα πράγματα που αποδείχθηκαν λανθασμένα. Και ο λόγος που γίνεται η ρύθμιση είναι ότι ο προϋπολογισμός πλέον θα πρέπει να προσαρμοστεί σχετικά με το κομμάτι της ανάθεσης έργων και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτός ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ το 2016. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κάποια ενδιαφέροντα θέματα για τους διαγωνισμούς που αφορούν σε μικρότερες προθεσμίες, ηλεκτρονική ανάθεση, ευελιξία ή τη δυνατότητα της εκτονιστέρων των τροποποίησης συμβολέων που κατακυρώθηκαν μέσω διαγωνισμών. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε, να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε. Αυτή λοιπόν η μεταρρύθμιση είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί ίσως να πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία να τροποποιήσουμε κάποια πράγματα σε αυτή τη δεκαετία. Γιατί δεν έχω την εντύπωση ότι η Κομισιόν ε, θέλει να αλλάζει συνεχώς ε, τον κανονισμό, περί, τον δημοσιονομικό κανονισμό. Ούτε κι εγώ. Πάντως, θα ε, επεξεργαστούμε τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης. Έχει ήδη συσταθεί η σχετική ομάδα εργασίας και σε τεχνικό επίπεδο ξεκινήσαμε τις ε, διαπραγματεύσεις και τις συνεδριάσεις το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Βεβαίως θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία από τη στιγμή που θα υπάρχει πολιτική συμφωνία επί του κειμένου. Και υπάρχει, υπάρχουν δύο εξαιρέσει. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Ελέγχου Προπλογισμών θα γνωμοδοτήσουν. Εγώ την περιμένω εναγωνίω περιμένουν αγωνίως και τις δύο αυτές γνωμοδοτήσεις. Βεβαίως ε, πρέπει να σας πω ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους και ισχύουν και για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Παρ' όλα αυτά εμείς ε, Κάναμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ζωή των υπαλλήλων στον ε, τομέα των εξωτερικών υποθέσεων. Περιμένω αναγωνίως τέλο πάντων τι θα κατατεθεί. Στις 3 Δεκεμβρίου θα καταθέσω το σχέδιο της έκθεσής μου και μέχρι τι 8 Ιανουαρίου του 2015 έχετε χρόνο να καταθέσετε τροποποίηση. Η ψηφοφορία θα είναι στις 5 Φεβρουαρίου και μετά θα ακολουθήσουν οι διαπραγματεύσεις ε, στο πλαίσιο του Τριμερού διαλόγου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι τροπολογίε, αλλά να είστε και λιγάκι προσεκτικοί όσον αφορά τη δημιουργικότητά σας. Ε, δεν ξέρω αν ε, θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα. Ξέρετε, το λέω αυτό γιατί έχω κάνει τόσο δυσάρεστη εμπειρία με τροπολογίες που δυστυχώς είμαι αναγκασμένη να το πω αυτό που είπα. Όσον αφορά λοιπόν την τράπεζα δεδομένων, η Transparency International διατύπωσε πέντε σημεία κριτικής που θα τα δω πολύ προσεκτικά, να δω κατά πόσον κάποια από αυτά μπορώ να τα υιοθετήσω. Εμένα αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια εύρυθμα λειτουργούσα τράπεζα δεδομένων. Όχι δηλαδή να ε, μπλεκόμαστε σε πάρα πολλά πράγματα που τελικά δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και είμαστε αναγκασμένοι να αποτύχουμε. Η τράπεζα δεδομένων να είναι αποτελεσματική. Και όπως σας είπα, μέχρι τώρα η εμπειρία μου δεν ήταν θετική. Εκτός λοιπόν από την τράπεζα δεδομένων, έχω και εγώ να καταθέσω κάποιες ε, τροπολογίες στο 108, στο υπαριθμό 5, εκεί που γίνεται λόγος για την υποχρέωση των κρατών μελών να ενημερώνουν τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με για λόγους αποκλεισμού από κάποιον διαγωνισμό. Μετά, στα ΣΔΙΤ, στα ΣΔΙΤ υπάρχει, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια κοινή δήλωση. Public private partnerships. Αυτή την κοινή δήλωση θα τη συμπεριλάβουμε διότι ε, νομίζω ότι ε, πρέπει να συμφωνήσω σε αυτό το τομέα. Κατόπιν υπάρχει και θα υπάρξει από μένα ένας ορισμός των διεθνών οργανισμών για ευνόητους λόγους. Γιατί ξέρετε, στον τομέα αυτό, αν δεν είμαι σαφής, θα εμφανιστούν άλλοι οργανισμοί που θα ισχυριστούν ότι είναι διεθνείς, ενώ δεν θα είναι. Και στην περίπτωση αυτή θα τους εκταμιευτούν κονδύλια χωρίς διαγωνισμούς. Υπήρξαν αυτές οι περιπτώσεις κατά το παρελθόν. Δέκα χρόνια ασχολούμαι το θέμα και έχω κάνει τη σχετική εμπειρία. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ε, θα είμαι πολύ πιο αυστηρή στον ορισμό του Διεθνής Οργανισμός. Κατόπιν η εσωτερική έλεγχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι ένα θέμα στο οποίο βρισκόμαστε σε διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτό θέλουμε να έχουμε καλύτερη ενημέρωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρίως για την απαλλαγή. Γιατί αν τελικά ως κοινοβούλιο δεν εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που μας προσφέρονται, αυτό είναι λάθος. Υπάρχουν και ειδικέ εκθέσεις του ε, ελεγκτικού συνεδρίου. Μέχρι τώρα ε, δημοσιεύονται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και επίσης ε, προχωράμε και εμείς πολύ αργά στην επεξεργασία των σφαλμάτων. Αυτή λοιπόν η αντιφατική διαδικασία θα πρέπει τουλάχιστον να επιταχυνθεί στις ε, έκτακτες εκθέσεις. Ίσως μπορούμε να το σκεφτούμε να τις καταργήσουμε πλήρως. Θα το συζητήσω αυτό με το Ελεγκτικό Συνέδριο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά την ετήσια έκθεση θα πρέπει να επιταχύνουμε την αντιφατική διαδικασία, όπως λέγεται, για να μπορούμε να απαντάμε ταχύτερα, με μεγαλύτερη ταχύτητα, σε προβλήματα που εμφανίζονται στον προϋπολογισμό. Όσον αφορά την απαλλαγή, αυτή πρέπει να πω είναι πηγή ανεξάντλητων εμπειριών. Βεβαίως και πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε το Συμβούλιο στη διαδικασία της απαλλαγής. Το έχουμε ε, δοκιμάσει αυτό επανειλημμένα. Κατόπιν υπάρχει και άλλο ένα θέμα το οποίο μας δημιουργεί όλο και περισσότερο προβλήματα. Δηλαδή διαπιστώνουμε ότι στα κράτη-μέλη εμφανίζονται πολιτικοί οικονομικού κλάδου οι οποίοι από επιχειρήσεις κάνουν πολιτική σταδιοδρομία. Και τι γίνεται, εμφανίζονται σε θέσεις όπου καλούνται να διαχειριστούν κοινοτικά κονδύλια. Όμως δεν παρετούνται από τις επιχειρήσεις τους, του αντίον εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σε αυτές. Εδώ λοιπόν πρέπει να τεθεί το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή την πηγή δυσφήμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κράτη-μέλη, αυτήν να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε και γι' αυτό εγώ είμαι ανοιχτή για όλους τους συναδέλφους που έχουν να καταθέσουν μια ιδέα και που θεωρούν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Ο πρόεδρος κύριος Γιούνκερ είπε ότι είναι η Επιτροπή της Έσχατης Ευκαιρίας, ίσως να είμαστε και το Κοινοβούλιο της Έσχατης Ευκαιρίας, τουλάχιστον όσον αφορά την διαχείριση των κονδυλίων. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της διαχείρισης των κονδυλίων. Είναι σημαντικό το τι ρυθμίζεται, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ενθαρρύνω τους νέους συναδέλφους, εφόσον ενδιαφέρονται, να έρθουν να συζητήσουν μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, θα καταθέσω την έκθεσή μου στις 3 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέσλε. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε εσά, το πρόσωπό σας για τον αγώνα κατά της απάτης και βεβαίως για την θέσπιση των βασικών αρχών μιας διοντολογίας την οποία πρέπει να τηρούμε. Μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στις 20 Ιανουαρίου και μετά 5 Φεβρουαρίου. Νομίζω αρκεί αυτό για την ώρα. Θα παρακαλέσω τον κύριο Σάρβαμα να αναπτύξει τώρα την έκθεσή του για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για έκθεση φιλανδικού ενδιαφέροντος για την παγκόσμια ναυτική, ναυτικό κλάδο δηλαδή, που έχει αντιμετωπίσει προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Οφείλω να πω ότι η Φιλανδία αντέδρασε με ταχύτητα και μάλιστα αρκετούς μήνες πριν υπέβαλαν, πριν να υποβάλουν αίτηση μάλλον, ξεκίνησαν προγράμματα και project. Μιλούμε για 600, 634 απολυμένους από το ναυπηγείο του Ράουα, ναυπηγείο του Ράουα στη Φιλανδία. Η επωνυμία του ναυπηγείου είναι STX και δραστηριοποιείται διεθνώς. σταμάτησαν τις δραστηριότητες τους και απέλησαν αυτά τα 634 άτομα. Λίγα στοιχεία από την έκθεσή μου έχουν ως εξής. Στην περιοχή του Τουρκού στη Φιλανδία, στην πόλη Ρώμα, κάνουν κάτι τι βεβαίως δεν είναι ρόλος του Κοινοβουλίου ούτε και δικό μου στόχος να δώσω μαθήματα στις χώρε μέλη. Ορισμένα πράγματα έχω περιλάβει ωστόσο στην εκθεσή μου με σκοπό να προσφέρω χείρα βοηθείας στους απολυμμένου για να βρουν δουλειά. Ο Δήμος της Ραούμα μας λέει ότι πιστεύει ότι θα μπορέσει να επανακατευθύνει και τον τελευταίο από αυτούς τους 634 σε νέες δουλειές. υπό την προϋπόθεση ότι τα σχέδιά τους θα ευοδοθούν, τα σχέδια του Δήμου δηλαδή. Οι άνθρωποι αυτοί, οι εργαζόμενοι αυτοί, οι απολυμμένοι εργαζόμενοι δηλαδή, είναι κάπως πιο ηλικιωμένοι, δεν έχουν πολλά προσόντα από άποψη εκπαίδευση και αυτό βέβαια αυξάνει τον κίνδυνο να μείνουν μακροχρόνια ανεργοί. Λοιπόν, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι ο σωστός παραλήπτης της αίτηση στην περίπτωση αυτή. Και γι' αυτό εγώ στηρίζω την αίτηση και αυτό περιλαμβάνω στην έκθεσή μου. Έχουμε, ρωτώ την γραμματεία, προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών. Υπάρχει ήδη. ο πρόεδρος. Δεν έχει μικρόφωνο ο πρόεδρος, τον ακούμε πολύ καλά. Τον ακούμε από το μικρόφωνο του κ. Σάρβαμα. Υπάρχει κάποια προθεσμία. 6 Νοεμβρίου. 6 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Δεν βλέπω ουδής να γύρει την χείρα για να λάβει το λόγο. Άρα, τα ξαναλέμε στις 20 Νοεμβρίου, όπου η Επιτροπή μας θα ψηφίσει. Η κυρία Γιάχτεν Μάκη, τώρα για την εταιρεία GAD στη Γαλλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην προκείμενη περίπτωση πρόκειται για μια γαλλική υπόθεση για μια επιχείρηση εγκατεστημένη στην Βρετάνη επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος που απέλησε, αναγκάστηκε να πωλήσει 720 άτομα. Η αιτιολόγηση της αίτηση που υποβάλλουν τώρα έχει ως εξής. Λέγουν ότι η κατανάλωση χείριου κρέατος έχει μειωθεί στη Γαλλία. Έχει κατέβει η κατανάλωση κιλών ανάτομο. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυξάνονται οι τιμές καταναλωτού για το χοιρινό κρέας. Αυξάνονται οι τιμές του χείριου κρέατος και έτσι δεν πάνε καλά τα πράγματα για την επιχείρηση. Αυτό ίσως έχει και κάποια σχέση με την παγκόσμια οικονομική κρίση. Βέβαια δεν είναι και αυτονόητη άμεση διασύνδεση, άμεση συνάφεια μεταξύ των δύο αυτών. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι δηλαδή που μειώνεται η κατανάλωση χοιρινού κρέατος στη Γαλλία, αλλά και αλλού. Αλλάζει και ο τρόπος ε, ζωής των ανθρώπων. Τώρα για την επιχείρηση αυτή μπαίνει και ένα θέμα κοινωνικού dumping μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και του στρεβλού ανταγωνισμού που οδήγησε σε επιδείνωση της θέσης της επιχείρησης αυτής μέσα στην κοινοτική αγορά. Ζητείτε λοιπόν με την γαλλική αίτηση 900.000 ευρώ για υποστήριξη προγραμμάτων για επανένταξη στην αγορά εργασίας των απολυθέντων. Θέλουν να φτιάξουν ένα είδος παροχής συμβουλών σε ένα one-stop shop για τους απολυμμένους εργαζόμενους. Θα αναλάβουν το έργο αυτό δε δύο επιχειρήσεις παροχής συμβουλών, δύο consulting δηλαδή, που είναι γνωστά τα ονόματά τους, εν προκειμένου, και αυτές θα λάβουν χρήματα βεβαίως από αυτό το ποσό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η αίτηση που έχει υποβάλει η Γαλλική Δημοκρατία εν προκειμένου πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι μπορούν να καταβληθούν οι 900.000 ευρώ. Έχει λάβει μεγάλη απήχηση το θέμα στη Γαλλία και έτσι εγώ τίνω να υποστηρίξω την θετική πρόταση της Κομισιόν. Σας ευχαριστούμε κυρία Γιατερμάκη. Οι τροπολογίες για την έκθεσή σας ε, μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 12 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας έχει προβλεφθεί για τις 20 Νοεμβρίου. Στην έκθεση αυτή φαίνεται η ανάγκη ε, σύγκλησης ε, και σε φορολογικά θέματα και σε θέματα εργατικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η έλλειψη σύγκλησης δημιουργεί τεράστιο κόστος. Επίσης, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να ενεργοποιείται σχετικά έγκαιρα και όχι κατόπιν εορτής αφού έχουν στο μεταξύ συντελεστεί απολύσεις. Καλό θα ήταν να αποτρέπονται οι απολύσεις με την κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Περάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Η πρώτη μας ψηφοφορία είναι ενδεικτική ψηφοφορία, γιατί δεν έχουμε ακόμη τη θέση του Συμβουλίου και αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2014. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 3, 4, 5, 6 και 7. Είναι ένα σύνολο. Όλοι αυτοί οι προϋπολογισμοί συνιστούν ένα πακέτο ο εισηγητής ο κ. Δεπρέ. Θα πρέπει να προσθέσουμε και την κινητοποίηση του αποθεματικού για πρόβλεπτες ανάγκες για το 2014 στο πακέτο μας. Συνδυάζεται με τον διορθωτικό προϋπολογισμό, προϋπολογισμό υπαριθμό 3. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή δεν χρειάζεται. Στις 20 Νοεμβρίου θα επανέλθουμε στο θέμα του αποθεματικού για τις απρόβλεπτες ανάγκες. Ωραία. Ποιοι είναι υπέρ των σχεδίων διορθωτικού προϋπολογισμού. Πρόκειται για ένα πακέτο που απαρτίζεται από τους προϋπολογισμούς 3, 4, 5, 6 και 7. Κατά. Ουδής. Αποχές. Τρεις αποχές. Περνάμε τώρα στις τροπολογίες της έκθεσης Στέφανετς ε, για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την περίπτωση Άντερσεν της Ιρλανδίας. Για την παράγραφο 1. Ποιος είναι υπέρ, ο εισηγητής είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Κανείς. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Τροπολογία 2. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Τρεις κατά. Δύο αποχές. Εγκρίνεται και η τροπολογία αυτή. Παραγράφος 7.1. Τροπολογία 3. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Ο εισηγητή είναι υπέρ. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται στην παράγραφο 7β, τροπολογία 4, ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7 σε. Τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11α. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ κατά, τρεις κατά, αποχές καμία, εγκρίνεται η τροπολογία. Παράγραφος 12, τροπολογία 7, ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά, χωρίς αποχές, 12β, τροπολογία 8, ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά, αποχές, Δύο αποχές χωρί αρνητικέ ψήφου εγκρίνεται. Τροπολογία 9 για την παράγραφο 12. Ο γιατί είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Δύο. απόχέ, καμία. Εγκρίνεται. Περνάμε στην παράγραφο 13α, τροπολογία 10. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Χωρίς αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο της έκθεσης ε, όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Le scrutin Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με 25 ψήφους υπέρ, 3 κατά και καμία αποχή. Ψηφίσουμε τώρα τις τροπολογίες της έκθεσης Νεγκρέσκου για την περίπτωση Sprider Stores στην Ελλάδα. Παράγραφος 2, τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ, ο εισηγητής είναι υπέρ. Κατά, Εγκρίνεται. Για την παράγραφο 2.1, τροπολογία 2. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. 3. κατά, χωρίς αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 3. Προφορική τροπολογία του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, καμία. Τροπολογία 5, τροπολογία 4, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 6, τροπολογία 5, ο εισηγητής είναι υπέρ, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, 6β, τροπολογία 6, ο εισηγητής είναι υπέρ, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, δύο αποχές, τρει ψηφοι κατά, 6C. Τροπολογία 7. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Τρει ψήφοι κατά, αποχές, καμία, εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Τροπολογία 8. Προφορική τροπολογία του εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Τροπολογία 9. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Καμία. Καμία αποχή. 9α. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Χωρίς αρνητικές ψήφους και χωρίς αποχές. Εγκρίνεται. 9β. Τροπολογία 11. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δύο, τέσσερις ψήφοι Εγκρίνεται. Τροπολογία 12, παράγραφος 10. Ποιος είναι... Α, έχει καταπέσει, συγγνώμη. 10α, α, τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ, ο εισηγητής είναι υπέρ. Κατά. Τρεις ψηφικάτα. κατά. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ και 3 κατά. Χωρίς αποχές. Τώρα, τμήμα 3. Προϋπολογισμός 2014. Έκθεση ΔΕΠΡΕ. Ο εισηγητής παρακαλώ. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι να περάσουμε στην ψηφοφορία για τις μεταφορές 34 και 35. Είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των προϋπολογισμών που μόλις υπερψηφίσαμε. Ζητώ λοιπόν από τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν τις δύο μεταφορές πιστώσεων 34 και 35. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Τρεις ψήφοι αποχές, καμία. Εγκρίνονται. Λοιπά τμήματα. Προϋπολογισμός 2014. Ή μάλλον προηγουμένως ε, ε, καταστάσεις προσωπικού της Επιτροπής και της Όλαφ. Κύριε Πρόεδρε, στην προηγούμενη συνεδρίαση και απενεργοποιείτε το μικρόφωνο του κύριου Ντεπρέ. Συγγνώμη. Στη προηγούμενη συνεδρίαση είχα ζητήσει από τους συναδέλφους να μην δεχτούμε αμέσως τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητήσαμε συμπληρωματικές αιτιολογήσεις ε, για να στοιχειοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αιτήματά της. Είναι ικανοποιητικές οι πληροφορίες και η ενημέρωση που λάβαμε. Γι' αυτό σας στείλω να υπερψηφίσουμε τις δύο τροποποιήσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ε, καταστάσεις καταλόγων. Ποιος είναι υπέρ των δύο τροποποιήσεων για την Κομισιόν και την ΟΛΑΦ. Ευχαριστώ. Κατά κανείς, καμία αποχή. Ωραία, εγκρίνεται. Πάμε στα λοιπά τμήματα. Ο κύριος Φερνάντες αντικαθιστά σήμερα την κυρία Χολμάιερ. Μας έπεισαν οι εξηγήσει, έπεισαν την εισηγητριά μας, την κυρία Χολμάιερ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους τη κυρίας Χολμάιερ θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι κατά των τριών ε, μεταφορών πιστώσεων. Στην Επιτροπή Περιφερειών ενισχύεται η δημοσιονομική γραμμή ε, για την επίσημη εφημερίδα, για την ε, κινητικότητα στις μεταφορές. Είναι απαραίτητες ε, οι μεταφορές αυτές για τις δημοσιεύσεις και για να βελτιωθεί η κινητικότητα. Δεν, είμαστε, δεν είναι κατά των μεταφορών. Τώρα για το ελεκτικό συνέδριο. 200.000 ευρώ είναι το προτινόμενο ποσό για τους μισθούς. Για να πληρωθούν οι μισθοί. Και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η μεταφορά πιστώσεων στόχο έχει την κάλυψη των μισθολογικών αναπροσαρμογών. 4,6 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό και θα πρέπει να ενισχυθούν και κάποιες δημοσιονομικές γραμμές σημαντικές. Η εισηγήτρια σας προτείνει η υπερψήφιση των τριών μεταφορών πιστώσεων. Σας ευχαριστούμε κύριε Φερνάντες για την αντικατάσταση της ηγετρίας. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί τις τρεις μεταφορές. Ωραία. Ψηφίζουμε από κοινού λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ των τριών μεταφορών πιστώσεων. Κατά. Αποχές. Δύο αποχές. Εγκρίνονται οι προτάσεις. Ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία. Υπάρχει κάτι για τα διάφορα μήπως. Όχι. Αυτά λοιπόν, λύεται η συνεδρίαση. Παρακαλώ τους συντονιστές να παραμείνουν στην αίθουσα, γιατί σε τρία λεπτά θα ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών.